Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάμε λοιπόν με την αποστηματινή μα συνεδρίαση και χαίρομαι που μπορώ να καλωσορίσω σήμερα εδώ μαζί μα τον νέο πρωθυπουργό, νέο πρωθυπουργό τη Μορδαβία, Πάβελ Φίλιπ. Τα θερμά μα συγχαρητήρια, κύριε Φίλιπ, για την εκλογή σα στο αξιώμα σα. Συνοδεύεται από την πολυάλμα... Χαλουβίτση, την πρόεδρο της Βουλής και την Βαλετίνα Χαλουβίγα την επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Μολδαβίας και αποτελεί προφανώς η Μολδαβία ένα σημαντικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς μία από τις λίγες χώρες με την οποία έχουμε μία Έχουμε συμφωνήσει μια συμφωνία εμπορίου και έχουμε ήδη μια εταιρική σχέση και βρισκόμαστε ήδη στην πρώτη, στο πρώτο, στην πρώτη χρονιά της εφαρμογής αυτών των συμφωνιών και πάντοτε ως κοινοβούλιο εμείς υποστηρίζαμε την ευρωπαϊκή προοπτική της ε, Μολδαβίας. Γνωρίζουμε όμως ταυτόχρονα ότι η Μολδαβία βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση η οποία ασκείται από την πλευρά της Μόσχας. και μιλάμε για ένα άλλο είδος πίεσης από αυτό που ασκείται από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Είναι πιο εκλεπτισμένη αν θέλετε η πίεση που ασκείται στη Μολδαβία αλλά όχι λιγότερο επικίνδυνο. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο εσωτερικό της ε, Μολδαβίας. Δηλαδή δεν έχουν συντονιστεί ακόμα οι προευρωπαϊκές ε, δυνάμεις μετά από την τελευταία συνάντηση του ευθυνοπόρου. Ελπίζουμε όμω πως αυτή η νέα κυβέρνηση τώρα της Μολδαβίας θα μπορέσει να αποφύγει τις πρόορες εκλογές, θα μπορέσει να ολοκληρώσει κανονικά την πολιτική της θητεία. και θα μπορέσει να εξασφαλίσει μια σταθερότητα χωρίς να χρειαστεί δηλαδή μέσω νέων εκλογών να ξεκινήσει και πάλι ε, το έργο της. και εκείνοι οι οποίοι θεώρησαν πως δεν ήταν ενδεδειγμένο να συμμετάσχουν στην ε, κυβέρνηση λόγων και των όσων ε, συνέβησαν κάτω το τελευταίο έτος και την καθαίρεση δηλαδή της προηγούμενης ε, κυβέρνησης να πω ότι θα ήθελα τώρα μέσα σε αυτήν τη νέα συντηρία να αναδειχθούν οι προευρωπαϊκές δυνάμεις. Θεωρώ σημαντικό τα σημαντικά βήματα τα οποία μας υποσχεθήκατε σε ό,τι αφορά για παράδειγμα ε, την υιοθέτηση του νομοθεσίας για την εισαγγελία θα εφαρμοστούν στην πράξη και ελπίζουμε να σημειωθεί και το πρόοδο σε σχέση με τα διάφορα νομοθετικά πακέτα, για παράδειγμα στον τομέα της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα θέλαμε επίσης να ακούσουμε κάτι από εσάς σε σχέση με την απόφαση του συνταγματικού σας δικαστηρίου της 4ης ε, Μαρτίου ότι δηλαδή οι προεδρικές εκλογές ε, θα λάβουν ε, χώρα μέσω του δημοψηφίσματος και να μας πείτε δηλαδή κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι σκόπιμο κατά τη δική σας άποψη παρότι βέβαια το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι μάλλον συμπολικό δεν έχει δηλαδή ε, ιδιαίτερα εκτεταμένη εξουσία. Σα δίνω όμω ε, τώρα το λόγο κύριε Πρωθυπουργέ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο Μπροκ που μου έδωσε την ευκαιρία αυτή να έρθω σήμερα και να παρουσιάσω στην Επιτροπή σας τις προτεραιότητες της κυβέρνησης της Μολδαβίας. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στηρίζει και αντιμετωπίζει φιλικά την Μολδαβία και τους κατοίκους της και αυτό το έχει αποδείξει πολλές φορές μέχρι τώρα. Έχει φανεί αυτό από τις ψηφοφορίες που έχετε κάνει και τις τοποθετήσεις σας στην Ολομέλεια. Τον Νοέμβριο του 2014, για παράδειγμα, όπου επικυρώθηκε η Συμφωνία Σύνθεσης και όταν ε, άνοιξαν ορθάνυχτα οι πόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους κατοίκους της Μολδαβίας ώστε να μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς την υποχρέωση θεώρησης. Η Μολδαβία συμφωνεί με το αναφέρονται στο κεφάλαιο 49, στο 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μολδαβία όμως φαίνεται να έχει τιμωρηθεί για την επιλογή που έκανε προς ε, τον ευρωπαϊκό δρόμο. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια παράγοντες ε, οι οποίοι έχουν επηρεάσει την επιλογή μας αυτή. Όντως τα γεγονότα μας έχουν επηρεάσει αρνητικά, όμως οι ευρωβουλευτές σας ανεξαρτήτως εποδίων ξέρουν ότι θέλουμε να προχωρήσουμε στο σωστό δρόμο. Είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και να οδηγηθούμε σε θετικές αλλαγές στις ζωές των πολιτών μας. Θέλουμε να εφαρμόσουμε τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου και Συναλλαγών, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ε, μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε και τους θεσμούς μας. ανέλαβα την Πρωθυπουργία σε μια περίοδο που θα ήταν πιο εύκολο να αφήσω κάποιον άλλον να αναλάβει τα ενία της χώρας. Όμως, με την κυβέρνηση δεχτήκαμε την ευθύνη αυτή. Αναλάβαμε δηλαδή την ευθύνη για σφάλματα που έγιναν κατά το παρελθόν, αλλά και για όσα θέλουμε να πετύχουμε στο μέλλον. Σκοπεύουμε να μην αφήσουμε τις συγκυρίες να υπερισχύσουν και να μας επιβληθούν. Θέλουμε να είμαστε κυβέρνηση η οποία θα επιστρέψει την Μολδαβία στο σωστό δρόμο προκειμένου να σταθεί στα πόδια της. Χτες είχαμε την δεύτερη συνάντηση του Συμβουλίου Σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Μολδαβία. Κατά τη διάρκεια αυτού του Συμβουλίου συναντήθηκα με την είπα το εκπρόσωπο Μοκερίνη και συζητήσαμε για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης. Το Συμβούλιο μας ε, παρουσίασε κάτι σαν δοκιμή προκειμένου να μπορούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε αποτελέσματα. Αγαπητοί φίλοι, θα σας παρουσιάσω τώρα τις προτεραιότητες της κυβέρνησής μας για φέτος. Στη συνέχεια θα αναφερθώ σε συγκεκριμένες δράσεις που αναλάβαμε από τότε που αναλάβαμε την κυβέρνηση και τρίτον θα σας μεταφέρω κάποιες σκέψεις μου για το πώς βλέπω τις εξελίξεις της σχέσης της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτεραιότητες της κυβέρνησής μας πρώτα απ' όλα είναι σαφείς και συνοψίζονται σε τρεις στόχους. Θέλουμε να διασφαλίσουμε πολιτική σταθερότητα και πραγματικό διάλογο ανάμεσα στην κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών. Θέλουμε να διασφαλίσουμε μακροοικονομική σταθερότητα υπογράφοντας συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ενίσχυση συνεργασίας με όλους τους εταίρους μας και εφαρμογή δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Πριν από λίγο καιρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας συζήτησε μαζί μας για το κατά πόσο θα έπρεπε να υπάρξουν πιο αυστηρά μέτρα όπως το ψήφισμα του Ιανουαρίου του 2016 για το DCFTA όσον αφορά τις σχέσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Νομίζω ότι οι προτερότητες της κυβέρνησης είναι κάτι που πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία των πολιτών και η αντιπολίτευση, αλλά και όλοι μας οι εταίροι. Θέλω να σας διασφαλίσω για τις προτερότητές μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Και η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Υπάρχει συμφωνία στην πλειοψηφία στη χώρα μου ότι οι μεταρρυθμίσεις για την χώρα είναι αναγκαίες. Πρέπει να προσφορήσουμε και εμείς το κοινοτικό εκτιμένο προκειμένου να καταφέρουμε περισσότερα. Ακόμα και η αντιπολίτευση στη Βουλή δεν έχει αντίρρηση γι' αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι οι προτεραιότητες, το να τεθούν οι προτεραιότητες δεν είναι το πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολο είναι τα πράγματα που μένει να γίνουν. Είναι ξεκάθαρο ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν αμέσως, χωρίς καθυστέρηση. Αγαπητέ Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό για μας. Όταν θα έχουμε εφαρμόσει τους στόχους της μεταρρύθμισης των θεσμών του κράτους, πρέπει να φροντίσουμε και για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του κόσμου στους πολιτικούς και στη λειτουργία των, ε, της δικαιοσύνης και των δημοκρατικών θεσμών της χώρας. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο σημείο της παρουσίασής μου τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δηλαδή που έχει πετύχει σε 1,5 μήνα η κυβέρνησή μας, από τότε δηλαδή που ανέλαβε καθήκοντα. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την πολιτική σταθερότητα, η κυβέρνηση αυτή έχει μια σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα και είναι πρόθυμη να ακολουθήσει το δρόμο που έχει καθορίσει η κυβέρνηση στα πλαίσια και τη Συμφωνία Σύνδεσης. Από τις πρώτες κιόλας μέρες φροντίσαμε να ηρεμήσει η πολιτική ζωή και είχαμε την ευκαιρία να έχουμε διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Οι ισχυρισμοί και οι διαμαρτυρίες ελήφθησαν υπόψη στον καθορισμό του προγράμματός μας. Η παρέτηση του Γενικού Εισαγγελέα, η έγκριση νόμων ακυρεότητας και η ανεξαρτησία των ρυθμιστών στο τραπεζικό τομέα ήταν κάτι που εγώ προσωπικά ήθελα να προχωρήσω, γιατί έχω την πεποίθηση πως η κοινωνία των πολιτών πρέπει να ελέγχει το τι συμβαίνει στην πολιτική ζωή. Η κοινωνία των πολιτών στην Μολδαβία μπορεί και πρέπει να αποτελεί μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και πρέπει να μπορεί να πιέζει την κυβέρνηση. Νομικά λοιπόν διαθέτουμε τους μηχανισμούς ώστε να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών στη διαδικασία αυτή αποφάσεων, ήδη από την αρχή από το σχεδιασμό των νόμων και η κυβέρνηση και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτήν την σχέση η οποία πρέπει να είναι μόνιμη. Ένας από τους στόχους μας λοιπόν είναι να μεταρρυθμίσουμε τους υπάρχοντες μηχανισμούς έτσι ώστε να συμμετέχει σε σταθερή βάση η κοινωνία των πολιτών σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Τώρα στα πλαίσια της συμφωνίας σύνδεσης βασιζόμαστε πολύ στην ε, ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών. Θέλουμε να μπορεί να ελέγχει και να εκφράζει απόψεις όσον αφορά τα διάφορα στοιχεία της συμφωνίας αυτής σύνδεσης. Οι εκπρόσωποι της Μολδαβίας στην πλατφόρμα αυτή πρέπει να μπορούν να κάνουν παρατηρήσεις και δηλώσεις για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Συμφωνία Σύνδεσης αναφέρθηκα και στην ανάκτηση εμπιστοσύνη του κόσμου. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πετύχουμε μόνο εφόσον έχουμε μια ανοιχτή στάση, εφόσον υπάρχει επικοινωνία και εφόσον συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών. Θέλουμε να ενισχύσουμε και να παγιώσουμε αυτήν την καλή σχέση με την κοινωνία των πολιτών. Οργανώνουμε λοιπόν ειδικέ συνεδριάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου με εκτελεστικές επιτροπές από την κοινωνία των πολιτών και στις διάφορες περιφέρειες, στην Ουκούσια και αλλού. Είχαμε και δράσεις στα πλαίσια ομάδας εργασίας με αυτονομίες όσον αφορά την αυτονομία ακριβώ της Ουρκόζια θέλουμε να προωθήσουμε μια στρατηγική μέθοδο για τις μειονότητες οι οποίες θα μπορούν μεταξύ άλλων να προωθήσουν την ποικιλομορφία στην κοινωνία και να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή. Θέλουμε να διευκολύνουμε δηλαδή το διαπολιτισμικό διάλογο. Μια άλλη διάσταση στην οποία επικεντρωθήκαμε τις 8 εβδομάδες που είμαστε στην κυβέρνηση είναι ισχυροί θεσμοί και αυτό για να πετύχουμε τους στόχους μας που είναι η ανεξαρτησία των θεσμών αυτών. Έτσι οθετήσαμε νομοθεσία ώστε οι θεσμοί να είναι ανεξάρτητοι όπως η δικαιοσύνη από την κυβέρνηση. Επίσης έχουμε νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης. Μειώσαμε από πέντε σε δύο τις άδειες που μπορεί να έχει ένα μόνο άτομο. Επίσης ασχολούμαστε με την προστασία των καταναλωτών, των περιβάλλων και άλλα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται και στη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου αλλά και τη Συμφωνία Σύνδεσης. Με τέτοιο γρήγορο ρυθμό λοιπόν καταφέραμε να, να κινητοποιήσουμε την πολιτική βούληση και έτσι να περάσουν νόμοι που οδηγούν σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Τον Φεβρουάριο είχαμε και μία αποστολή του Διεθνούς Μασοτικού Ταμείου που ήρθε για να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για μία νέα συμφωνία συνεργασίας. Από 1η Μαρτίου στείλαμε έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δράσεις που θέλουμε να εφαρμοστούν μέχρι τον Ιούλιο στη Μολδαβία λαμβάνοντας υπόψη και τους ισχυρισμούς της κοινωνίας των πολιτών. Είναι ένα έγγραφο το οποίο υπογράφει ο Πρωθυπουργό αλλά και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Αντικατοπτρίζει την ευθύνη που αναλαμβάνουν όλοι, η ευρεία πλατφόρμα δηλαδή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Τέλος, αγαπητοί ευρωβουλευτές, θέλω να σας παρουσιάσω τις δικές μου ιδέες για τις μελλοντικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας. Όπως έχω πει μέχρι τώρα, αυτά που πρέπει να κάνουμε, που μένει να κάνουμε, είναι ξεκάθαρα. Και είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντική για να πετύχουν οι προσπάθειες που κάνουμε για μεταρρυθμίσεις. Η πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος στόχος των σχέσεών μας. Είναι ένας στόχος ο οποίος ελπίζω ότι θα καταλήξει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Εγώ δεν έρχομαι εδώ να σας ζητήσω επιταγή εν λευκό. Όχι. Ξέρω ότι η εμπιστοσύνη κερδίζεται. Αυτή είναι η δικιά μου αντίληψη και η αντίληψή μας στη Μολδαβία. Λαμβάνοντα υπόψη και την απόφαση του δογματικού Δικαστηρίου που συνάδει με τις δικές μας προσδοκίες για πολιτική σταθερότητα, Πρέπει να ομολογήσω ότι για μένα προσωπικά όταν λήφθη η απόφαση αυτή εξεπλάγει. Δεν νομίζω ότι κάποιος που είναι Πρωθυπουργό θέλει να έχει προεκλογική εκστρατεία για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Συγχρόνως όμως είμαι πεπισμένος ότι αυτή η απόφαση βασίζεται και σε σημαντικά επιχειρήματα. Από την άλλη προσπαθώ να βρω και τις θετικές πτυχές. Προεδρικές εκλογές στην Μολδαβία με κοινοβουλευτική στήριξη είναι κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική κρίση. Γιατί δεν πετυχαίνουμε πάντα να έχουμε αρκετές ψήφους στο Κοινοβούλιο. Αν έχουμε απευθείας εκλογές για τον Πρόεδρο, αυτό θα σημάνει σίγουρα ότι θα εκλεγεί ο πρόεδρος και ότι δεν θα οδηγηθούμε σε κρίση ή σε περιορισμούς που θα οδηγήσουν σε πρόορες εκλογές στη συνέχεια. Ζήτησα λοιπόν από όλα τα μέλη της κυβέρνησή μου να μην συμμετάσχουν πολύ στην προεκλογική εκστρατεία και να αποφύγουν δηλώσεις ως εκτελεστική εξουσία πρέπει να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένες δράσεις που είναι και ο κανονικός μας ρόλος. Είμαι στη διαθεσή σας τώρα αν έχετε ερωτήσεις και ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε έναν ανοιχτό και επικοδομητικό διάλογο. Προηγουμένως όμως θέλω να σας πω ότι η πλειοψηφία μας είναι αποφασισμένη χωρίς καθυστέρηση να θέσει εφαρμογή τις μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν την ζωή των πολιτών μας και θα βοηθήσουν να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη τους σε εμά. Η Συμφωνία Ελεύθερου Αμπορίου αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για να επιτεθεί ο στόχος αυτός. Ε, σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Πρωθυπουργέ. Έχουμε λοιπόν τώρα κάποιους ομιλητές. Θέλω να πάρω το λόγο. Κύριος Πρέντερ. Εκπλήσουμε που είναι ο πρώτος, αλλά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζω εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω και έναν άλλο συμμετέχοντα όμως, ο οποίος ε, η οποία ήταν σχεδόν πρωθυπουργό, αλλά ο δικό συνασπισμό την απέρριψε. Επειδή είχε πει ότι θα καταπολεμούσε τη διαφθορά, αν δεν κάνω λάθο. Το πρώτο μου ερώτημα έχει λοιπόν να κάνει με αυτό ακριβώ το ζήτημα. Τι κάνετε εσεί για τη διαφθορά, για ποιο λόγο θεωρείστε εσείς πιο αξιόπιστο για τον κυβερνώντα αυτό συνασπισμό και για ποιο λόγο εσεί θα καταφέρετε να καταπολεμήσετε καλύτερα τη διαφθορά. Ένας προκάτοχός σας που είχε έρθει εδώ πέρα στο παρελθόν δεν είχε καταφέρει να μας δώσει μία απάντηση αξιόπιστη. Τι κάνετε εσείς όμως προκειμένου να καταφέρετε να γλιτώσετε από την επιρροή που έχει ο κύριος Πλαχώτινεν, ο ολιγάρχης αυτός, ο σημαντικός επιχειρηματίας της Μολδαβίας είναι πάρα πολύ σημαντικό στο μέλλον να μην επηρεάζει την πολιτική κατάσταση και τις πολιτικές εξελίξεις αυτός ο ολιγάρχης. Όσον αφορά τώρα τα θεσμικά όργανα της ε, Μολδαβίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτά να ανεξάρτητα και να μην επηρεάζονται και να μην ελέγχονται από τους ολιγάρχες. Ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστώ. κύριε Πρωθυπουργέ. σα ευχαριστώ που είσαστε σήμερα εδώ. Είχαμε κάνει ούτως ή άλλως και μία διμερή ε, συνάντηση στο παρελθόν και είχαμε κάνει ένα οικοδομητικό διάλογο. Προφανώ η Μολδαβία είναι μια σημαντική διαλογο Προφανώ η μολδαβια ειναι μια σημαντικη χωρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δούμε τα όσα έχουν λάβει χώρα ε, στην ε, Μολδαβία μέσα στα τελευταία δύο χρόνια θα διαπιστώσει ότι έχουν γίνει πολλά. Για παράδειγμα, πρόοδο σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, ζώνη ελεύθερων συναλλαγών εταιρική σχέση. Και ταυτόχρονα βέβαια η Μολδαβία αποτελεί ε, μια χώρα η οποία λαμβάνει τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κεφαλήν. Άρα λοιπόν βλέπουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει όσα πραγματικά μπορούσε ε, προ όφελο τη Μολδαβία και θα συνεχίσει να το πράττει και στο μέλλον. Η σταθερότητα, η πολιτική σταθερότητα είναι απολύτω απαραίτητη. Προφανώ αυτό είναι σαφέ, αλλά είναι απαραίτητη και για να μπορέσετε να επιτύχετε κάποια πρόοδο και έχετε θέσει τώρα κάποια θεμέλια. Για παράδειγμα η νέα νομοθεσία η οποία έχει ήδη ψηφιστεί από το ε, από τη Βουλή σας. Ε, πράγματι αυτό το νομοθετικό λοιπόν πακέτο θα πρέπει τώρα να εφαρμοστεί στην πράξη και αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι είναι δύσκολο το έργο σας. Ε, βρίσκεστε σε ένα μονόδρομο. Δεν μπορείτε δηλαδή να, έχετε, να ακολουθήσετε κάποια ένα άλλη εναλλακτική. Μόνο προς τα μπροστά μπορείτε να πάτε. Ε, θα κλείσω όμως λέγοντας ότι πραγματικά θα πρέπει να θέσετε σε ύψιστη προτεραιότητα του ε, τους ίδιους τους ανθρώπους, τους πολίτες σας. Και αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμόσετε το ταχύτερο δυνατόν την ε, σχέση σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο έχετε συμφωνήσει με την Επιτροπή. Σα καλώ λοιπόν να το τηρήσετε. Thank you, Chair. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, ξέρετε ότι στο παρελθόν σε μια συνάντηση στο Κισινάου ενημερωθήκαμε για τα φαινόμενα διαφθοράς και για αυτή την απίστευτη περίπτωση διαφθοράς, το τεράστιο αυτό ποσό το οποίο εξαφανίστηκε, υπεξαιρέθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Τι πρόκειται να κάνετε για να αποφύγετε ανάλογα φαινόμενα διαφθοράς στο μέλλον και προκειμένου να μην έχουμε πλέον περιπτώσεις ατιμορρησίας για τέτοια εγκλήματα. Πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά επίσης το ζήτημα της ασφάλειας για την υπερνηστερία. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Thank ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά τις υφιστάμενες σχέσεις σας με την Ουκρανία. Υπάρχουν ε, περιπτώσεις συνεργασίας στα σύνορά σας. Επίσης, τι κάνετε με τα σύνορα που έχετε με την υπερθνιστερία. Επίσης, πιο συγκεκριμένο όσον αφορά την υπερθνιστερία. Επί του παρόντος υπάρχει κάποιο σχέδιο επανενσωμάτωσης της υπερθνιστερίας στην Μολδαβία ή προβλέπετε κάτι τέτοιο για το μέλλον. Γιατί πριν από μερικά χρόνια είχαν γίνει κάποιες απόπειρες, κάποιες προσπάθειες για την επίλυση της διένεξης, αλλά είναι πολύ σημαντικό και στο μέλλον, εφόσον το μέλλον σας προβλέπει μια ευρωπαϊκή προοπτική, να καταφέρετε να επιλύσετε το πρόβλημα το οποίο υφίσταται ακόμα με την υπερνηστερία. Ähm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πριν από μερικές εβδομάδες ε, με δύο συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισκέφθηκα το Κισινό και ε, πρέπει να πω ότι τρομοκρατήθηκα λίγο από τις ε, συνομιλίες που έκανα εκεί. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς προσωπικά, ο σχηματισμός της τελευταίας κυβέρνησης είναι αποδεκτός κατά τη γνώμη σας, γιατί ειδικότερα οι φιλοευρωπαϊκοί πολίτες ε, που συνομίλησαν μαζί μας ε, μας είπαν ότι αυτή η διαδικασία του συμμετισμού της σημερινής κυβέρνησης ήταν εντελώς αντιδημοκρατική. Μετά σε ό,τι αφορά αυτό το σκάνδαλο της ε, υπεξαίρεσης του αιώνα πραγματικά ε, ε εξετάσετε εδώ και πολύ καιρό. Τι έχει συμβεί, θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι. είναι, έχουν εμπλακεί ευρωπαϊκές τράπεζες σε αυτό το σκάνδαλο. Μπορείτε επίσης να μας πείτε κατά πόσο θα ήσασταν διατεθειμένος να συμμετάσχει η Eurojust στη διαλεύκανση αυτού του σκανδάλου. Και εν πάση περιπτώσει μπορείτε να μας δώσετε κάποιες κάποια νέα σε σχέση με τη διαλεύκανσή του. Γιατί βέβαια ε, υπήρξε μια πολύ βαριά κατηγορία η οποία ε, ε, διαφάνηκε σε όλες τις συζητήσεις που κάναμε από μερικές εβδομάδες. Δηλαδή μας είπαν οι εκπρόσωποι ότι ναι είμαστε φιλοευρωπαϊκοί, είμαστε φιλοευρωπαϊστές, αλλά αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε μια τόσο μεγάλη διαφθορά. Σήμερα το πρωί άκουσα ότι το συνταγματικό, δικαστήριο της Μολδαβίας έχει ε, μεταβάλει τις ε, προϋποθέσεις για τις προεδρικές εκλογές, ότι δηλαδή θα είναι δυνατή τώρα πλέον η άμεση εκλογή του Προέδρου, όπως ήταν δηλαδή δυνατό πριν από το 2001. Ταυτόχρονα όμως άλλαξαν και οι προϋποθέσεις της υποψηφιότητας, για να μπορέσει δηλαδή κάποιος να δεθεί υποψήφιος ως Πρόεδρος. Δηλαδή θα πρέπει να έχει ζήσει για συγκεκριμένο αριθμό χρόνων ως πολίτης της Μολδαβίας, εντός της Μολδαβίας και θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη ηλικία από 40 ετών. Τι είναι αυτό, δεν παρεμβαίνετε ε, με κάποιο τρόπο στη συνταγματική διαδικασία και δεν ε, ουσιαστικά αποδεικνύεται ε, πραγματική κατηγορία ότι δηλαδή υπάρχει ανάμειξη πολιτική στις συνταγματικές διαδικασίες της χώρας και ότι δεν λειτουργούν δηλαδή σωστά τα θεσμικά όργανα. Κύριε Πρωθυπουργέ, καταρχάς να πω το εξής. Είχα πάει στον Ταμπάσα και θεωρώ ότι ε, η περιοχή αυτή ανήκε στο παρελθόν στη Ρωσία, δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο για τη Μολδαβία. Η Μολδαβία έχει ένα δυτικό παρελθόν, ανήκει στη Δυτική Ευρώπη και γενικότερα γίνανε προσπάθειες ε, και από τους τσάρους ε, να καταφέρουν σιγά σιγά να την προσαρτήσουν στο ρωσικό έδαφος, στη ρωσική αυτοκρατορία. Καταλαβαίνω βέβαια ότι εσείς ανήκετε ή θέλετε να ανήκετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να τηρήσετε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ισχύουν βέβαια και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφάνεια, χρηστή διαχείριση κτλ. Νομίζω ότι από αυτού πρέπει να σημειωθεί ακόμα σημαντική πρόοδος. Αυτό που ήθελα να τονίσω και θεωρώ, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό προκειμένου να καταφέρετε να συμβάλλετε σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποτελέσετε ένα είδος γέφυρας. Εγώ, όντας, αλσατός, θεωρώ ότι θα πρέπει να γεφυρώνουμε τις διαφορές μας. Θα πρέπει να γεφυρώσετε κι εσείς τις διαφορές που έχετε αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία. Η Ρωσία υφίσταται, αποτελεί τμήμα της Ευρώπης και νομίζω ότι το χειρότερο που θα μπορούσατε να κάνετε είναι να επιλέξετε να κάνετε αυτό που έκανε η Ουκρανία, δηλαδή να επιλέξετε μία ρήξη με τη Ρωσία, να αποτελέσετε σύνορο, να αποτελέσετε τείχος και να μην αποτελέσετε γέφυρα. Βλέπετε αυτή τη στιγμή πως οδηγήθηκε σε αποτυχία η Ουκρανία και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να καταβάλει το αντίτιμο. Θεωρώ ότι θα καταφέρει τελικά στο τέλος ε, η Ρωσία να υποφεληθεί από την κατάσταση αυτή. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας ότι ε, κλείνεται περισσότερο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλα αυτά είναι σημαντικό στα πλαίσια της μεγάλης αυτής Ευρώπης να αποτελέσετε μια γέφυρα με τη Ρωσία και σας καλώ επίσης να κρατήσετε ουδέτερη στάση απέναντι στο ΝΑΤΟ γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρετε να κατευνάσετε τις διενέξεις που υφίστανται ακόμα στην περιοχή σας. Ah, ναι, η Front National μας είπε, μας είπε δηλαδή ότι η Μολδαβία για παράδειγμα ανήκει στη Ρωσία και ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουμε σταθερότητα. Εν πάση περίπτωση. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ, νομίζω πως ε, το ζητούμενο εδώ είναι αυτό το οποίο ανέφεραν ήδη κάποιοι συνάδελφοι, δηλαδή ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν οι πολίτες της Μολδαβίας να έχουν εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα του κράτους. Δεν θα πρέπει δηλαδή να έχουν την εντύπωση ότι απλά πρόκειται για ένα παραπέτασμα πίσω από το οποίο υπάρχουν άλλοι οι οποίοι κινούν τα νήματα. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να καταστεί σαφές, να υπάρχει διαφάνεια για τους πολίτες και αναφέρθηκε βέβαια και σε αυτό το πλαίσιο και το μεγάλο σκάνδαλο το οποίο πλήττει ε, τη χώρα σας αυτή την περίοδο και με την εξαφάνιση αυτού του τόσο μεγάλου ποσού. Θα ήθελα λοιπόν σχετικά με αυτό το ζήτημα να σας θέσω ένα ερώτημα. Τίθεται γενικότερα αυτό το ερώτημα, δηλαδή σε ποιον ανήκουν τελικά τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας. Ε, κάτι τέτοιο, εάν θα μπορούσατε δηλαδή να το ξεκαθαρίσει αυτό, θα αποτελούσε και μια μεγάλη ε, συμβολή για τη διαφάνεια. Δηλαδή να υπήρχε τελικά μια δημοσίευση των στοιχείων ιδιοκτησίας των ε, τραπεζών της ε, Μολδαβίας. Και τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή σε επίπεδο περάκτων εταιρεών. Όσο. Ε, τώρα αναφερθήκατε στο ότι θα υπάρξουν νέες ρυθμίσεις στον οπτικο-ακουστικό τομέα και από τις πέντε άδειε τώρα να άτομα έχουμε ε, πάει στις δύο. Όμως ε, ε, σας εξηγώ ότι η αποκέντρωση την οποία θέλετε να επιτύχετε ενδεχομένως δεν θα είναι δυνατή αν κινηθείτε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πώς θέλετε να έχετε μία απεμπλοκή από τα συμφέροντα του οπτικοακουστικού τομέα με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης ε, θα ήθελα ε, να μου πείτε τι θεωρείτε πως συμβαίνει στο επίπεδο των δραστηριοτήτων που έχει αναλάβει η ε, Ρωσία. Δηλαδή τα φιλορωσικά κόμματα και το γεγονός ότι έχουν τόσο ε, μεγάλη επιρροή μέσα στην πολιτική ζωή της Μολδαβίας αποτελεί απλά και μόνο ένδειξη ότι τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα δεν έχουν καταδείξει ε, την αξία του τι ακριβώς δηλαδή θα μπορούσαν να κερδίσουν οι πολίτες της Μολδαβίας με μια ε, στενότερη σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Uh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα συνεχίσω μιλώντας την ε, ρουμανική γλώσσα, τη γλώσσα της Ρουμανίας και της ε, Μολδαβίας. Κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε ότι ε, η Μολδαβία μέσω της ιστορίας της, της γλώσσας της, της γεωγραφικής της θέσης ανήκει στην νοτιοανατολική Ευρώπη και όχι στην Ευρασία. Προφανώς εσείς θα πρέπει τώρα να εφαρμόσετε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς επίσης και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα όμως, αγαπητέ Πρωθυπουργέ, βλέπουμε ότι ε, η ρωσική προπαγάνδα του παρελθόντος αλλά και η σημερινή συνεχίζουν και διαδίδουν διάφορες φήμες. Αυτό το έχουμε δει όχι μόνο στη Μόσχα, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, αλλά ακόμα και στη Μολδαβία λένε ότι οι Μολδαβοί ουσιαστικά είναι σλαβωνικής καταγωγής, ενώ εμείς γνωρίζουμε ότι έχουν λατινική καταγωγή. Γνωρίζουμε ότι ανήκεται ουσιαστικά στην ιστορία του ρουμανικού λαού. Επίσης διαδίδονται διάφορες φήμες όσον αφορά την ε, ιστορία της όλης περιοχής που εμείς ονομάζουμε ε, Βαρσαραβία. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με όλα τα ζητήματα αυτά και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να καταπολεμήσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες παραπληροφόρησης που γίνονται για την ιστορία της Μολδαβίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω όχι μόνο να έχουμε κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις αλλά και μεταρρυθμίσεις στον εκπαιδευτικό τομέα παντού σε όλη την επικράτεια της ε, Μολδαβίας Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία δεν μπορούν να παρακολουθούν το σχολείο στη μητρική τους γλώσσα, δηλαδή τη ρουμανική γλώσσα. Αν οι πολίτε τη Μολδαβία δεν ξέρουν το παρελθόν του, δεν ξέρουν από πού προέρχονται, τότε δεν μπορούν να γνωρίζουν και πού θέλουν να κατευθυνθούν. Δεν είναι καλύτερο εσεί να του λέτε ότι ανήκουν πολύ περισσότερο στη Ρουμανία και κατ' επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στην Ευρασία. Γιατί ξέρετε ότι γίνεται μια πολύ εντατική προπαγάνδα αυτή τη στιγμή, ιδίω στην ύπεθρο τη Μολδαβία, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί υποστηρικτέ των Ρώσων οι οποίοι λένε ότι η διαβίωση των πολιτών, οι μισθοί και οι συντάξει του θα ήταν πολύ καλύτερε αν ανήκανε στην Ευρασία. Εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα αν έρθετε πιο κοντά σε εμά, στη Ρουμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you, Chair. Mr. Prime Minister. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα και εγώ να σα ε, καλωσορίσω από την πλευρά μου στι ε, Βρυξέλλε και την προσωπία σα μεταξύ άλλων και των προεξωτερικών σα αλλά και την μεγάλη αντιπροσωπεία από την Μολδαβική Βουλή. Νομίζω δηλαδή αυτή η εβδομάδα θα μπορούσε να ονομαστεί ω η εβδομάδα τη Μολδαβία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πράγματι εγώ πρέπει σε πολύ ανοιχτές και επικοδομητικέ συνομιλίε μαζί σας στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν δηλαδή συναντηθήκαμε στο Κισινάου και εντυπωσιάστηκα από την αποφασιστικότητά σας, δηλαδή να συνεχίσετε με τις ε, μεταρρυθμίσεις ε, που επιθυμούσατε. Θα πρέπει να σας πω βέβαια ότι ε, δεν ήσασταν πολύ αισιόδοξο τότε. Τώρα στις Βρυξέλλες εμφανίζεστε πολύ πιο θετικός, γιατί βλέπουμε πως ο σημερινός κυβερνητικό συνασπισμός είναι πιο πολλά υποσχόμενος και μας είπατε ότι ήδη έχετε εφαρμόσει κάποιες από αυτές τις μεταρρυθμίσεις, όχι όλες αλλά κάποιες από αυτές. Εγώ λοιπόν ε, χαιρετίζω το γεγονό ότι έχει ξεκινήσει και πάλι τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων Μολδαβία. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Σωστά υπόθηκε αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή ε, άλλο μέλλον για τη Μολδαβία πέρα από αυτό, πέρα από τη μεταρρύθμιση και ελπίζω το μέλλον της Μολδαβίας να είναι ευρωπαϊκό. Εκτιμώ τις ε, προσπάθειες που έχετε κάνει από την πλευρά σας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον οδικό χάρτη, ο οποίος έχει πλέον επολυθεί και είναι ε, επίσης σημαντικό ότι κάποια πράγματα ήδη έχουν επιτευχθεί. Για παράδειγμα η διοικητική μεταρρύθμιση, όπως ε, ο διορισμός ενός νέου διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, ε, νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εισαγγελία. Άρα λοιπόν θεωρώ θετικό το να εφαρμοστεί ταχύτερα, να εφαρμοστούν ταχύτερα αυτές οι μεταρρυθμίσεις από ό,τι προβλέπεται μέσα στου επομενου ενα ένα-δύο γιατί είμαστε εταίροι προφανώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μολδαβία. Όμω κύριε Πρωθυπουργέ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιστύχει μια συμφωνία Μολδαβία και με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Υπήρξε και μια προκαταρκτική αντιπροσωπεία του, του ε, στη Μολδαβία αλλά θα υπάρξει και μία νέα αντιπροσωπεία που θα επισκεφθεί την ε, ε, Μολδαβία για την ε, μία νέα συμφωνία. Οπότε θα ήθελα να μα πείτε κάτι σχετικά. Δηλαδή, ποιε είναι οι προοπτικέ σύναψη μία συμφωνία με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Ποιε είναι οι πιθανότητε θεωρείτε ότι υπάρχουν για τη σύναψη μια τέτοια συμφωνία. Γιατί βέβαια παρακολουθήσαμε τα όσα συμβαίνουν με κάποια απογοητεύση σε σχέση με αυτό το ζήτημα στη Μολδαβία και ελπίζουμε πω θα υπάρξει μια αλλαγή στο μέλλον σχέση με αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, θέλω να πω ότι σίγουρα υπάρχουν πολλά ωφέλη για τον λαό της Μολδαβίας αν υπάρχει προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση δεν είναι υπέρ της Ευρώπης μόνο όταν το λέει όμως, αλλά όταν εφαρμόζει τη Συμφωνία Σύνδεσης ανάμεσα στην Μολδαβία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημείωσα λοιπόν για το χάρτη πορείας όσον αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής σύνδεσης και το πρώτο σημείο είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς. Συγκεκριμένα όμως θέλω να σας ρωτήσω τι θα κάνετε για να βελτιώσετε τη λειτουργία της Επιτροπής ακεραιότητας και του Κέντρου κατά της διαφθοράς. Τι πρωτοβουλίες θα προτείνετε και πώς θα παρακολουθήσετε την εφαρμογή των μέτρων αυτών, γιατί η εφαρμογή είναι η ουσία. Όσον αφορά τώρα τις απάτες στο τραπεζικό τομέα, αναφέρθηκαν σε αυτό πολλοί συνάδελφοι. Εγώ νομίζω ότι τρία πρέπει να γίνουν. Πρώτον, να καλυφθούν τα χρήματα, οι απόλυες μέχρι την τελευταία δεκάρα. Έγιναν έρευνες, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχουν αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται και συνεργασία με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα οποία ίσως να έχουν περισσότερη εμπειρία όσον αφορά την, ε, τις απάτες, την νομιμοποίηση παρανομού χρήματος κλπ. Τι θα κάνετε λοιπόν για να ανακτήσετε τα ποσά αυτά, τι θα κάνετε για να συνεργαστείτε με άλλα θεσμικά όργανα και τι θα κάνετε για να ανακτήσετε την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών προκειμένου να επενδύσουν στη Μολδαβία και πώς θα εποπτεύσετε καλύτερα εφ' εξής στον τραπεζικό τομέα ώστε τέτοιες περιπτώσεις σαν και αυτή που είχατε να μην επαναληφθεί. Ωραία να υπάρχει κεντρική τράπεζα, διοικητής, ναι, αλλά η εποπτεία της ε, Κεντρικής Τράπεζας που πολιτικά είναι ανεξάρτητη πρέπει να υπάρχει ένας ε, νέος ε, διοικητής, δεν φτάνει και μπορείτε να μας δώσετε και κάποιες λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση της Μολδαβίας. Βλέπουμε ότι υπάρχει υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, ότι ο πληθωρισμός είναι πάρα πολύ ψηλός, υψηλότερος τα τελευταία 7 χρόνια και οι εξωτερικές επενδύσεις μειώνονται στην Μολδαβία. Τι θα κάνετε λοιπόν με όλους αυτούς τους δείκτες που επιδεινώνονται. Τα δημοσιονομικά επίσης της Μολδαβίας θα επιδεινωθούν στο μέλλον. Άρα δεν θα δημιουργούνται πια θέσεις απασχόλησης τους επόμενους μήνες στη Μολδαβία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο, ο Μποστινάρο. Κύριε Πρωθυπουργέ. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Δεν θέλω εδώ να τσακωθούμε το ΕΛΚΑ και οι σοσιαλιστές για το παρελθόν της Μολδαβίας, γιατί για να παραφράσω κάτι που λέμε στην Μολδαβία, αν υπάρχει διχασμός μεταξύ μας και οι δύο φταίμε. Και οι δύο πλευρές έχουν τις αδυναμίες και ο Πρωθυπουργό είναι από μια συγκεκριμένη πολιτική οικογένεια και έχει συνεισφέρει και αυτό στην ε, κρίση στη χώρα. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα για να βοηθήσουμε τη Μολδαβία. Και θέλω να πω και στους συναδέλφους ότι δεν υπάρχει καμία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να ενδιαφέρεται περισσότερο για την ακαιρεότητα της Μολδαβίας από τη Ρουμανία. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν καλά όλοι οι συνάδελφοι. Να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Τώρα για αυτά που έχετε δεσμευτεί να κάνετε. Ε, μίλησαν και οι συνάδελφοι για τον χάρτη πορείας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Η νομοθεσία για την Κεντρική Τράπεζα και τις αρμοδιότητές της και τα κριτήρια για την επιλογή του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Πότε θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Δεύτερον, αναφέρθηκε η τεράστια απάτη. Τεράστια για το μέγεθος της Μολδαβίας. Πότε θα έχουμε κάποια ελάχιστα τουλάχιστον αποτελέσματα της έρευνας για το τεράστιο αυτό σκάνδαλο. Το πήγε σαν αποτέλεσμα να χάσει την εμπιστοσύνη του ο κόσμος στα πολιτικά κόμματα και τους θεσμούς. Τρίτη ερώτηση. Πολλοί στη Μολδαβία μιλούν για επιθετική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων που απειλεί τελικά την ε, ίδια την ασφάλεια της Μολδαβίας. Η κυβέρνησή σας τι θα κάνει για να μην υπάρχουν κίνδυνοι ασφάλειας που έχουν να κάνουν ε, με αυτό τον υβριδικό πόλεμο που τόσο καλά γνωρίζουμε στην Ευρώπη και που πολλοί από εμά δεν θέλουν να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει. Και τέλος, σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Και όχι λόγω πολιτικής οικογένειας, αλλά γιατί τίθεται θέμα πρόωρων εκλογών. Όσοι πιστεύουν σε αυτήν την ψευδέστηση, ορεινά το ότι και οι σοσιαλιστές θα κερδίσουν, που καταγγέλουν τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και ρεαλιστές για το τι εξελίξεις θέλουμε στη Μολδαβία και να υποστηρίξουμε εσάς. Και να λάβουμε υπόψη μας ε, και τις διάφορες αποχρώσεις που έχουν αυτά τα ζητήματα και να μην είμαστε απόλυτοι. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, λέει η κυρία Νικολάη. Είμαι μία από αυτούς που χαίρεται που έχει κυβέρνηση η Μολδαβία υπό εσά και ελπίζω εσείς να είσαστε πράγματι ο Πρωθυπουργό της τελευταίας ευκαιρίας, γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία της Μολδαβίας. Αλλιώς θα είχαμε πρόορε εκλογές που θα ήταν καταστροφή για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας σας. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία. Έχω μία ερώτηση προς εσάς. οι επιπτώσεις της απόφασης του Σταγματικού Δικαστηρίου. Ως νομικός εκπλήσωμαι. Αλλά πρέπει να δεχτούμε την απόφαση ως έχει. Πότε αναμένετε τις προεδρικές εκλογές. Γιατί αυτό θα επηρεάσει και την ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις σας τις οποίες καλωσορίζω. Καλωσορίζω την αποφασιστικότητά σας για μεταρρυθμίσεις. Έχετε σκεφτεί τι επιπτώσεις θα έχει η εκλογή Προέδρου στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος. Γιατί οι Ρουμάνοι ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Πρέπει να στηρίζεται από όλες τις πλευρές η ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Τόκες. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως εκπρόσωπος της Ουγγρικής μειονότητας και ως πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου της Ουγγαρίας στην Τρασιλβανία, θέλω να σας εκφράσω την υποστήριξή μας. Υποστηρίζουμε τον αγώνα σας κατά της διαφθοράς. Ως Πρωθυπουργός αποτελείται την τελευταία ευκαιρία για τη δημοκρατία της Μολδαβίας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι για τη ρουμανική ταυτότητα σε αντιπαράθεση με την ε, μολδαβική ταυτότητα. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι η Σερβία αμφισβητεί τη ρουμανική ταυτότητα ορισμένων ή ότι η Ρωσία δεν αναγνωρίζει την ρουμανική ταυτότητα πολιτών που ζουν στη Μολδαβία. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα. Σύμφωνα με διάφορα ενωτικά κινήματα στη Μολδαβία, σας αντιμετωπίζουν πραγματικοί Ρουμάνοι. Κάτι το οποίο διευκολύνει τις δικές μας δραστηριότητε και τις δικές μας προσπάθειες να σας υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο στις προσπάθειές σας προσέγγισης με την Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο ιστορικά, αλλά και για το μέλλον να συνεχίσετε στην πορεία αυτή της εθνικής ενότητας. Και ακόμα και αν ζούμε σε δύο διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Και να σας ρωτήσω και κάτι για τις μειονότητες στην ε, Μολδαβία. Για μας τους Ούγκρους είναι ένα παράδειγμα η αυτονομία των Γαγκάρων. Πώς πάνε τα πράγματα στην κακοσία λοιπόν και ποια είναι η κατάσταση των ρωσόφωνων μειονοτήτων στη Μολδαβία. Και κάτι ακόμα για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ξέρω ότι υπάρχει διάσπαση μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σας ρωτάω, μια που και ίδιος είμαι κληρικός. Ένα τμήμα είναι πιο κοντά στην Ρωσία, το άλλο είναι πιο κοντά στη Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Η διάσπαση αυτή, αυτό το σχίσμα, τι ρόλο παίζει, τι επιπτώσεις έχει πάνω στην εθνική ενότητα της Μολδαβίας. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος, δυστυχώς. Αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, καταρχά να σε ευχαριστήσω. Να σε ευχαριστήσω για όλε αυτέ τι παρατηρήσει για όλε αυτέ τι ερωτήσει που θέσατε. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντήσω. Να απαντήσω τις περισσότερες τουλάχιστον από τις ερωτήσεις σας, με τη σειρά που τις άκουσα. Καταρχάς, θα ήθελα να επαναλάβω ότι και εγώ ίδιος, αλλά και το σύνολο της κυβέρνησής μου, συνειδητοποιούμε πλήρως πώς έχουν τα πράγματα στη δημοκρατία της Μολδαβίας. Γνωρίζουμε πώς έχει η κατάσταση και έχουμε αντλήσει διδάγματα από το παρελθόν. Γνωρίζουμε πλέον ποια είναι τα βαθύτερα αίτια της κρίσης. Και πραγματικά λυπούμεθα που απογοητεύσαμε και τους πολίτες της Μολδαβίας και τους ξένους εταίρους μας. Γι' αυτό το λόγο στην αρχική μου παρέμβαση είπα ότι ο βασικός στόχος της κυβέρνησης αυτής είναι να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας απέναντι στους πολίτες μας, απέναντι στα θεσμικά όργανα και απέναντι στην πολιτική τάξη. και ότι θέλουμε να ανακτήσουμε επίση και την εμπιστοσύνη των ξένων εταίρων μα, προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο την ευρωπαϊκή πορεία τη Μολδαβία. Και όταν μιλάω για ευρωπαϊκή πορεία, ειλικρινά γνωρίζω, γνωρίζω πολύ καλά πώ έχουν τα πράγματα. Δεν κάνω εδώ απλέ δηλώσει, προσπαθώντα να πείσω τον έναν τον άλλον. Θα ήθελα πραγματικά να με κρίνετε με βάση τις πράξεις μου και με βάση τα αποτελέσματα των πράξεών μου. Και θα ήθελα εδώ πέρα ανοίγοντας με παρένθεση να κάνω την εξής έκκληση. Μη μας κρίνετε με βάση τα όσα γίνανε στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν. Νομίζω ότι θα πρέπει αν είμαστε ένα δέντρο για παράδειγμα, αν ναι, μας κρίνετε με βάση τις ρίζες μας που ουσιαστικά έχουν να κάνουν ε, με το πρόσφατο παρελθόν της χώρας και τις αποφάσεις προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά με βάση τους καρπούς που θα, θα παράξουμε. Τώρα όσον αφορά την ε, επιρροή των ολιγαρχών, έγινε ε, από κάποιον μία αναφορά σε ορισμένα άτομα. και ανήκουν πολλές φορές στο ίδιο πολιτικό κόμμα με μάσα. Εγώ θεωρώ ότι η εναλλαγή των κομμάτων ή των πολιτικών δεν αλλάζει αναγκαστικά την κατάσταση της διαφθοράς. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Τα προβλήματα μπορούν να επιληθούν μέσω συστηματικής δράσης και ποιοτικών συστηματικών τροποποιήσεων του ίδιου του πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα έλεγα ότι στα πλαίσια του διακυβερνητικού μας συστήματος προσπαθούμε να αποφύγουμε τη χρησιμοποίηση γενικών όρων που θα οδηγούσαν σε καιροσκοπία. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι οργανώνουμε πλέον τις πολιτικές μας δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο στη Μολδαβία που θα μπορούμε πλέον να δίνουμε τις κατάλληλες λύσεις στην κατάλληλη στιγμή. Και να θέσω τα πράγματα και κάπως διαφορετικά. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία των πολιτικών κομμάτων προκειμένου να μην περιπέσουν στα λάθη του παρελθόντος, όπου ορισμένα μονοάτομα, συγκεκριμένοι πολιτικοί, επηρέαζαν όλη την πολιτική κατάσταση στη Μολδαβία εμείς εντοπίσαμε ως ε, λύση καταρχάς τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικές ομάδες στη Μολδαβία. Αυτό σαφώς μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ τη λειτουργία των κομμάτων και στο σχέδιο προπολογισμού για το 2016 προβλέπουμε πλέον τους αναγκαίους πόρους για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και ρυθμίζουμε πλέον τη χρηματοδότηση αυτή με τρόπο πολύ πιο ανοιχτό και αυστηρό. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν τα πολιτικά κόμματα τελικά να είναι ανεξάρτητα. Δεν θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να εξαρτώνται από ένα ή περισσότερα άτομα, γιατί τότε πραγματικά μπορούμε να μιλάμε όντω για επιρροή ολιγαρχών και κατ' επέκταση επιρροή των ολιγαρχών στην κρατική διακυβέρνηση. Θα ήθελα τώρα να περάσω σε κάποιες άλλες παρατηρήσεις και θα ήθελα να αφαιρθώ στον τρόπο με τον οποίο ανέλαβε την εξουσία η κυβέρνησή μου, το Υπουργικό Αυτοσυμβούλιο. Τα πράγματα μπορεί να μην εξελίχθηκαν πάρα πολύ ομαλά, πάντως σε κάθε περίπτωση αναλάβαμε την εξουσία τηρώντας πλήρως τα όσα λέει το Σύνταγμα της χώρας μου και είχαμε την υποστήριξη 57 μελών του Κοινοβουλίου και κατά αυτόν τον τρόπο επιταχύναμε την όλη διαδικασία ορκομοσίας και ξεκίνησε κατά αυτόν τον τρόπο η λειτουργία της κυβέρνησης. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε και κάποιες επικρίσεις για το έργο που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Επίσης, όσον αφορά την υπερνηστερία και όσον αφορά τις σχέσεις που έχουμε με την Ουκρανία. Κύριε Βανόρντεν, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Βανόρντεν, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Βανόρντεν, σας καλώ στην τάξη. Κύριε Βανόρντεν, ησυχία παρακαλώ. Όσον αφορά λοιπόν την υπερθνιστερία και όσον αφορά τη σχέση μας με την Ουκρανία, Εδώ θεωρώ ότι έχουμε κάποιες σημαντικές ε, ευκαιρίες. Η Γερμανία επί του παρόντος έχει την προεδρία του ΟΑΣΕ και είχαμε μια συνάντηση με την προεδρία λοιπόν του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας για την Ευρώπη και θεωρώ ότι μπορούμε μέσω κάποιων μικρών αλλά σημαντικών πράξεων οδηγηθούμε σε ένα βιώσιμο αποτέλεσμα. Μέχρι τα τέλη του Απριλίου προβλέπονται διαπραγματεύσεις με σύνθεση 3 συν 2 και μέχρι τα τέλη Μαΐου θέλουμε να έχουμε διαπραγματεύσεις με σύνθεση 5 συν 2. Όσον αφορά τώρα τις σχέσεις μας με την Ουκρανία, έχουμε ένα σχέδιο κοινών συνόρων όσον αφορά τη συνεργασία αστυνομικών και τελωνιακών δυνάμεων βρίσκεται σε φάση συζήτησης το πρόγραμμα αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει να ευοδοθεί και κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια πολύ καλύτερη συνεργασία με την Ουκρανία. Όσον αφορά τον τελωνιακό έλεγχο, θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως το πρόγραμμα αυτό και στη συνέχεια, όταν καλύψουμε όλα τα τελωνιακά ζητήματα, θα πρέπει να προχωρήσουμε και στη συνεργασία της συνοριοφυλακής αυτό θα είναι πάρα πολύ θετικό και για τους ε, ανθρώπους εκείνους που ζουν στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνίστερου και που δεν θα χρειάζεται κάθε φορά να περνάνε από το Κισινάου προκειμένου να εκτελονίζουν προϊόντα, αλλά θα μπορούν αυτό να το κάνουν επιτόπου. Όσον αφορά τώρα το σταγματικό δικαστήριο. Αναφέρθηκα στην αρχική μου παρέμβαση στο ζήτημα αυτό, θα επανέλθω όμως γιατί πολλοί θέσατε σχετικά ερωτήματα. Η απόφαση η οποία λήφθη... Βασίστε πάνω σε συγκεκριμένα επιχειρήματα. Έχουμε πει ότι εμείς στην κυβέρνηση θα προσπαθήσουμε να μην εμπλακούμε σε καμία περίπτωση στην εκλογική διαδικασία, αλλά θα επιτελέσουμε τις αρμοδιότητες προβλέπονται στα πλαίσια της εκτελεστικής εξουσίας. Η άμεση εκλογή Προέδρου από τους πολίτες έχει και κάποιες θετικές πτυχές είναι κάτι το οποίο ζήτησαν οι ίδιοι οι πολίτες της Μολδαβίας όταν με ένα ποσοστό άνω του 90% τάχθηκαν υπέρ των άμεσων εκλογών για τη θέση του Προέδρου. Θεωρούμε λοιπόν ότι από τις 23 Μαρτίου θα έχουμε μπροστά μας δύο μήνες μέχρι να λήξει η θητεία του υφιστάμενου Προέδρου και θα μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο μέσα σε αυτή τη δίμηνη περίοδο να καθορίσουμε και την ημερομηνία των προεδρικών εκλογών. Σε αυτή λοιπόν τη δίμηνη περίοδο θα πρέπει να προσαρμοστεί η εθνική μας νομοθεσία διότι όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή θα περάσουμε σε ένα νέο τρόπο εκλογής του Προέδρου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δώσουμε τα απαραίτητα στοιχεία και τους απαραίτητου πόρους σε αυτή τη νέα διαδικασία και να δώσουμε τα απαραίτητα στοιχεία και ενημέρωση στου πολίτε. Πρέπει επίσης να δούμε και ποιοι θα είναι οι πιθανοί υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου, ποιοι θα πάρουν το χρήσμα για τις προεδρικές αυτές εκλογές. Και είναι πολύ σημαντικό στη συνέχεια να επιτρέψουμε μια περίοδο 60 ή 90 ημερών για την εκλογική εκστρατεία. Αν κάνουμε τους υπολογισμούς, συνειδητοποιούμε ότι οι προεδρικές εκλογές θα γίνουν μάλλον τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Ενδεχομένω αυτή να μην είναι πλέον κατάλληλη περίοδο για προεδρικέ εκλογέ, αυτή τουλάχιστον η προσωπική μου γνώμη. Πάντω σε κάθε περίπτωση δεν θα λάβω εγώ την οριστική απόφαση, αλλά το Κοινοβούλιο της Μολδαβία, Σε κάθε περίπτωση οι εκλογές ενδεχομένως να γίνουν το φθινόπωρο, στις αρχές του φθινοπόρου. Τώρα, όσον αφορά ένα άλλο ζήτημα το οποίο εθίγει πολλές φορές από τους ευρωβουλευτές, ξέρετε ότι ε, μία αντιπροσωπεία εξεταστική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήρθε πρόσφατα στο Κισινάου. Πρέπει να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα και πέρα από κάθε πιθανή διαφορετική ερμηνεία ότι είχαμε πολύ επικοδομητικές συνεδριάσεις και επαφές με τους εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτή τη φορά δεν ετέθησαν καθόλου προϋποθέσεις στις σχέσεις μεταξύ Κισινάου και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν ετέθησαν νέες προϋποθέσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ασχοληθήκαμε κυρίως με την περίπτωση τριών τραπεζών που βρίσκονται υπό ειδική εποπτεία. Για δύο από αυτές έχει γίνει ήδη πλήρης έλεγχος και στα τέλη Μαρτίου θα ολοκληρωθεί και ο, ο, και ο της τρίτης τράπεζας και στην Ουάσιγκτον στη συνέχεια θα γίνει και μια συνεδρίαση μεταξύ εκπροσώπων της Μολδαβίας, του Υπουργού Οικονομικών συγκεκριμένα, και εκπροσώπων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στη συνέχεια ελπίζουμε μέσα σε ένα μήνα να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια οριστική επίσημη συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα, κατά πάση πιθανότητα, στις αρχές Ιουνίου θα έχουμε υπογράψει μια συμφωνία με τον Διεθνή Αυτό Οργανισμό. Δεν είναι αυτός σκοπό μα να καταφέρουμε να πάρουμε οικονομικού πόρου από το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Αν καταφέρουμε όμω να υπογράψουμε με τον οργανισμό αυτό μία συμφωνία, τότε θα έχουμε διαφορετικέ μορφέ χρηματοδότηση με του διεθνού μα εταίρου. Τώρα όσον αφορά τον οδικό χάρτη, ζήτημα το οποίο ετέθη από διάφορου συναδέλφου, επρόκειτο για μια πρωτοβουλία του Επιτρόπου Χάν, την οποία εμεί δεχτήκαμε πολύ θετικά. Ο δικός αυτό χάρτη αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και πρέπει να αναλάβει στο μέλλον η Δημοκρατία της Μολδαβίας σε σχέση με την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης. Ο δικός αυτός χάρτης προβλέπει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και για κάθε ξεχωριστή δράση προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες εφαρμογής. Εμείς σε κάθε περίπτωση έχουμε πει, προσωπικά το έχω πει ο ίδιος αλλά και πολλοί συναδελφοί μου, ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτόν τον οδικό χάρτη. Ξέρετε ότι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές της χώρας μου εξέτασαν ενδελεχώς τον οδικό αυτό χάρτη και χαρήκαμε πάρα πολύ όταν είδαμε ότι η πλειοψηφία των βουλευτών στο κοινοβούλιο της χώρας μου αποφάσισαν ότι θα πρέπει να εγκριθεί αυτός ο δικός χάρτης με την τροποποίηση βέβαια κάποιων προθεσμιών προκειμένου να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις επιμέρους δράσεις που βρίσκονται σε αυτόν τον δικό χάρτη. Όλοι όμως οι εκπρόσωποι στο Κοινοβούλιο συνειδητοποιούν τη σημασία αυτού του δικού χάρτη και συνειδητοποιούν πόσο σημαντικό είναι με τη βοήθεια των Βρυξελών να ολοκληρωθεί αυτός ο χάρτης και να εφαρμοστεί πλήρως. Ξεκινήσαμε λοιπόν ήδη κάποιε συζητήσεις και νομίζω ότι η συνεργασία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ επικοδομητική και με τους εκπροσώπους της Γκακαουζία. Ξεκίνησε ένας διάλογος ανάμεσα στους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου μας και τους εκπροσώπους της Λαϊκής Συνέλευσης της Γκακαουζίας και σε εκτελεστικό επίπεδο. Πρέπει να σας πω επίσης ότι στις 4 Μαρτίου διοργανώσαμε μία συνέλευση του Υπουργικού Συμβουλίου στην περιοχή της Γκακαουζίας και αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε σε κάποια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη αυτή περιφέρεια της Μολδαβίας και αυτό στη συνέχεια μεταφράστηκε σε συγκεκριμένες δράσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Δημιουργήσαμε μία μόνιμη επιτροπή η οποία μέσα σε ένα μήνα θα πρέπει να εντοπίσει όλα τα εκρεμή προβληματικά ζητήματα που έχουμε στην περιφέρεια της Γκακαουζίας και στη συνέχεια η επιτροπή αυτή θα προτείνει ένα, ένα κοινό σχέδιο δράσης το οποίο θα εγκριθεί από την εκτελεστική εξουσία του Κισινάου και από την εκτελεστική επιτροπή της περιοχής της Γκαγκαουζίας. Όσον αφορά την κοινωνία των πολιτών, ανέκαθεν ήμουνα υπέρ του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών. Ανέκαθεν αυτή ήταν η βασική μου πεποίθηση, ότι ανα πάσα στιγμή θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο ενδελεχής έλεγχος, η συνεχής παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου που θα προέρχεται από την κοινωνία των πολιτών. Και στο παρελθόν, όταν ήμουν απλός υπουργό, θεωρούσα ότι η πίεση που μας ασκεί η κοινωνία των πολιτών αποτελεί πραγματικό επικοδομητικό κίνητρο για ένα καλύτερο κυβερνητικό έργο. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι ως Πρωθυπουργό καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να έχουμε έναν συνεχή επικοδομητικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Ήδη έχουν γίνει πάρα πολλές συναντήσεις με πάρα πολλές ομάδες που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και έχουμε συζητήσει διάφορα ζητήματα. Ορισμένα από αυτά ήδη τα έχουμε επιλύσει και μαζί με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου θέλουμε να θεσπίσουμε ένα εθνικό συμβούλιο συμμετοχής στο οποίο θα εκπροσωπείται και η κοινωνία των πολιτών και θα υπάρχει μάλιστα και μια κοινή γραμματεία που θα καλύπτει το έργο της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών να μπορούν να εξετάζουν διάφορα νομοσχέδια ή να κάνουν επικοδομητικές προτάσεις όσον αφορά την προεξέταση στο κοινοβούλιο μας νομοσχέδια. Όσον αφορά τώρα το τραπεζικό και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Μολδαβίας, σίγουρα η τεράστια αυτή απάτη που έλαβε χώρα πρόσφατα ανατάραξε όλο το πολιτικό καθεστώς στην Μολδαβία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στο μέλλον διασφαλιστεί το έργο των θεσμικών οργάνων της χώρας προκειμένου να εντοπιστούν όλοι οι πέτοι, όλοι οι πέτοι της σημαντικότητας αυτής υπεξαίρεσης. Από την άλλη θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να καταφέρουμε να ανακτήσουμε τα χρήματα αυτά τα οποία υπεξαιρέθηκαν. Και κάτι ακόμα πιο σημαντικό είναι πολύ σημαντικό να δούμε σε ποιες δράσεις προχώρησαν οι αρχές της Μολδαβίας προκειμένου να μην επαναληφθεί τέτοια πάτη ποτέ στο μέλλον. Από τη μία λοιπόν πλευρά θέλουμε να ενδυναμώσουμε τους διάφορους ρυθμιστικούς ε, φορείς και φορείς όπως η Εθνική Επιτροπή για τις Χρηματοπιστωτικές Αγορές, καθώς επίσης να ενισχύσουμε και την ίδια την Κεντρική Τράπεζα της Μολδαβίας. Ήδη έχουμε γκρίνει νομοσχέδιο το οποίο αυξάνει τις αρμοδιότητες και την εξουσία των φορέων αυτών. Από την άλλη, προχωρήσαμε και στον διορισμό του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Μολδαβίας, εγκρίθηκε ο νέος αυτός διοικητής με απόλυτη διαφάνεια από το Κοινοβούλιο της χώρας μου και με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Χαίρομαι επίση πάρα πολύ για τη διαδικασία αυτή του διορισμού του διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα Μολδαβία συμμετείχε και ένα υψηλόβαθμο σύμβουλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε επίση, όπω σα είπα, ότι έγινε ένα ενδελεχή έλεγχος σε τρει συγκεκριμένε τράπεζε τη χώρα και είδαμε πραγματικά ότι μπορούμε να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα, μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε το τραπεζικό σύστημα και κατά αυτόν τον τρόπο να επαναφέρουμε μια κάποια σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας. Τέλος, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, όπως σας είπα στην αρχή της παρέμβασής μου, σας παρακαλώ πολύ, ας μας κρίνετε βάσει της δράσης μας. Ας μας κρίνετε βάσει των αποτελεσμάτων της δράσης μας. Η παρέμβασή μας, όλες οι αποφάσεις που λαμβάνουμε είναι απόλυτα δημόσιες. Εμείς θα σας κρατούμε ενήμερους για κάθε απόφαση που λαμβάνουμε και επιθυμούμε να έχουμε τη συμβολή και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, έγκριση του θεματολογίου σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μολδαβίας. Σας υπόσχομαι ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα στο σύντομο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Für die Zeit, die zur Verfügung standen. Σας ε, ευχαριστούμε εγκάρδια για τον χρόνο που διαθέσατε ε, για την επίσκεψή σας σήμερα εδώ και για τον διάλογο που κάναμε. Θεωρούμε πως θα αποτελέσει τη βάση για να, μια επικοδομητική συνεργασία μεταξύ μας, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και στις προσδοκίες των πολιτών της χώρας σας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο κύριε Πρωθυπουργέ. Thank you. Colleagues, let's start. Ας ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έχουμε στην εμερήσια διάταξή μας τις πληροφορίες σε αυτή τη φάση. Έχουμε ε, ζητήθηκε από τις συζητήσεις από την συγχύτρια κυρία Καλνιέτα και του σκιώδες συγκητής να αναβάλουμε τη σχετική ψηφοφορία και εγώ είμαι διατεθειμένος να το αποδεχτώ εφόσον όλοι σα συμφωνείτε και να καταγραφεί. Στα πρακτικό ότι θα τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει, δηλαδή ψηφοφορία τον Απρίλιο στην Ολομέλεια. Που σημαίνει φυσικά αυτό τι λιγότερο χρόνο για τι πολιτικέ ομάδε, δηλαδή προετοιμασία του εν ώψη τη ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Εάν δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει αντίρρηση θα αναβληθεί για την επόμενη εβδομάδα λοιπόν η ψηφοφορία για την ε, έκθεση της κυρίας Καλνιέτη. Και παρόλα αυτά η συζήτηση μετά η τελική και η ψηφοφορία θα γίνει τον Απρίλιο όπως έχει προβλεφθεί. Εάν λοιπόν συμφωνείτε όλοι περνάμε στην έκθεση της συγκεκριμένης κυρίας Πύρη Κύριε Πύρη, σα ε, δίνω με τελευταία ευκαιρία να πάρετε το λόγο, αν δεν θέλετε να τον πάρετε. Οπότε α ξεκινήσουμε κατευθείαν με την ψηφοφορία. οι 36, 39 και 174 έχουν αποσυρθεί εν λόγω τροπολογίες. Έτσι δεν είναι. Κύριε Βάλεβα. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα να γίνει ψηφοφορία επί των 36 και 39. Πρόεδρος. Όχι, έχουν αποσυρθεί οι τροπολογίες 36 και 39, οπότε δεν μπορούμε να ψηφίσουμε από αυτόν. Οπότε κλείσαμε αυτό το θέμα. Ποιος ε, χτυπάει εδώ παλαμάκια. παρακαλώ, το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να επισημάνω ότι αναφορικά με την τροπολογία μου 536 ε, η οποία αναφέρεται στον επικισμό των κατεχομένων εδαφών της πατρίδας μου της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία αντί να ενταχθεί τουλάχιστον στην παράγραφο 28α που, αναφέρεται στον ε, στον επικισμό έχει μπει κάτω από το Compromise 14 που αναφέρεται στο δίκαιο της θάλασσας. Αυτό είναι απαράδεκτο, το αντιλαμβάνεστε και αυτό ζητώ να γίνει ξεχωριστή ψηφοφορία στην τροπολογία μου 536 θα προβούμε ε, στην κανονική διαδικασία ψήφισης των συμβαστικών τροπολογιών όπως τις έχουμε μπροστά μας. Εδώ. Έτσι θα κινηθούμε. Και ε, ζητάτε και πάλι το λόγο, παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν, ότι παίρνουμε εμείς εκ μέρου μα τι τροπολογίε 36 και 39 και ζητάμε να ψηφιστούν. Αποσύρθηκαν, αλλά εμεί ω ομάδα τι αναλαμβάνουμε. Ω ομάδα 36 και 39 για να ψηφιστούν. Dann werden wir Καλώ, λέει ο πρόεδρο. Θα ψηφίσουμε λοιπόν επί των 36 και 39. Σύμφωνα με το άρθρο 169 παράγραφος 5 του καταστατικού μας. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Ναι, αναφέρεται λοιπόν στο σχετικό άρθρο ότι εάν αμέσω μετά την απόρριψη τη μια τροπολογία κάποιο άλλο αναλάβει την αλόγω ε, τροπολογία, τότε θα πρέπει να γίνει ψήφιση από αυτών των τροπολογιών. Αυτό προβλέπει λοιπόν το σχετικό άρθρο. Περνάμε στην ψηφοφορία. 101 ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τοπολογία 8. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όχι 100. Περνάμε στη συμβαστική τοπολογία 9. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 142 ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 183. Τροπολογία 183 σε τρία τμήματα. Τμήμα 1. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Hmm? We have to again. Πρέπει να ξαναρχίσουμε Ηλεκτρονική ψηφοφορία. <laughs> The vote is closed. Πέρασε η 39 ψήφοι υπέρ, 18 κατά, οπότε εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τη τροπολογία ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέσει, εγκρίνεται. Ψήφι, ε, τμήμα 3 ψήφι υπέρ. Α, όχι. Καταπίπτει το τρίτο τμήμα λόγω της συμβαστικής τροπολογίας 13. Οπότε περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 14. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 209. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 232. Τροπολογία 232. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 233. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 234 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. 234 λοιπόν ελέγχουμε. E Το ΕΛΚ ψηφίζει υπέρ τροπολογιών των σοσιαλιστών κατά ε, με την αντίθετη γνώμη των σοσιαλιστών. Σα ζητώ συγγνώμη αλλά με μπερδεύει αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Πέραση το ΕΛΚ λοιπόν κέρδισε, αν θέλετε, 36 ψήφοι υπέρ, 26 ψήφοι κατά. Συμβαστική τροπολογία 17 ψήφοι υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 245 ψήφοι υπέρ. Κατά. Ψήφι υπέρ ξανά. Δείξτε μου. Ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. 253 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 18 ψήφι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 265 ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται. 266 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 269 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 286 ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 288 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέραση της 43 ψήφοι υπέρ, 24 κατά εγκρίνεται. 290 ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 291 ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 302-303. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Θα ελέγξουμε. Πέραση ψηφοφορίας. 36 ψήφι υπέρ. 27 κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 20. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 συμβαστική, 21 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 304 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 305 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 308 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 307 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 309 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 310 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 311 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 312 υπέρ κατά ελέγχουμε πέρας της ψηφοφορίας ένας, ε, μια ψήφος παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, έλξη ψηφοφορία, 32 ψήφοι υπέρ, 34 κατά, οπότε απορρίπτεται. Περνάμε στην 313, αν δεν κάνω λάθος, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 314 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 306 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 330 τροπολογία σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 331 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 315 σε, στο δεύτερο τμήμα της ψήφι υπέρ του δεύτερου τμήματος. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 25 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται μαζί με την προφορική εδώ τροπολογία. Έτσι το oral amendment. Περνάμε στην συμβαστικό 27 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 28 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 378. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Πέραση της ψηφοφορίας. 35 ψήφοι υπέρ, 30 κατά, εγκρίνεται. 379. Λέει ο Πρόεδρος. Α, όχι, βιάστηκα λίγο, άρα έχουμε τη συμβαστική 29. Συμβαστική τροπολογία λοιπόν 29. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 379 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Ωραία, να ελέγξουμε. Πέραση της ψηφοφορίας. Συμβαστική τροπολογία 30 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 31 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 32 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απολογία 411. Συμπληρωματική. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 419 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 420 υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Ποιο φώναξε τσεκ έτσι τόσο πιστικά, λέει ο πρόεδρο. Έληξε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 421 υπέρ. Κατά. Ποιες απορρίπτεται. 422 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 423 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 424 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε. 424. try. 425 ψήφι πέρ Κατά. Αποχές. Και αυτή να την ελέγξουν Ενώ είμαστε σίγουροι. Λήξη της ψηφοφορίας. εδώ ίσα ίσα που υπερψηφίστηκε. Συμβαστική 33 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 438. Μόνο το δεύτερο τμήμα μου λένε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. θα ελέγξουμε. The vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Δεν ξέρω πια τι γίνεται, λέει ο πρόεδρος. Antrag 449-450. Τροπολογία 449-450 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 351 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 452 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 453 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε όμως Λήξη λοιπόν της ψηφοφορίας απορρίπτεται με 32 ψήφους υπέρ, 29 ε, κατά, συγγνώμη, 453 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. Πέραση της ψηφοφορίας. Αγκρίνεται. 38 εναντί 28. 356 ψήφοι υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 457 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 458 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 459 ψήφι υπέρ Α, όχι, καταπίπτει 459, οπότε πάμε στην 360 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 34. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 472 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Σε Συμβασική τοπολογία 34, λέει ο πρόεδρος. Four seven four. Where is in favor? 474. Ψήφι πέρα κατά αποχές απορρίπτεται. 473 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 475 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 476 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 477 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 478 υπέρ όχι, ξανά 477 ψήφι υπέρ. Τις 477 Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 478. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 479 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 480 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 481 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 482 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε τη 482. Λήξη της πληροφορίας. 37 ψήφοι υπέρ, 29 κατά, εγκρίνεται. 483 υπέρ, κατά, αποχές, καταπίπτει, ρωτάει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται, όχι, δεν καταπίπτει. 484 τώρα, ε, καταπίπτει. Οπότε 485 ψήφοι υπέρ. Κατά, αποχές, ελέγχουμε. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 487 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 488 ψήφι υπέρ. Κατά. «487 λοιπόν ξανά, ε, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 488 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 489 ψήφι υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Νομίζω πως απορρίπτεται. Πέρας της 29 ψήφι υπέρ, 38 κατά απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία ψήφι υπέρ, 35. Ε, κατά αποχές εκρίνεται 499 ψήφι υπέρ. 499, λοιπόν ψήφι υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Προδευτέρα ψήφι υπέρ, 26 κατά εγκρίνεται. Ε, Συγγείτε παίρνει το λόγο, είμαστε κατά της προφορικής τροπολογίας, της συμβιβαστικής τροπολογίας. Πρόεδρος, άρα τότε δεν είναι συμβαστική τροπολογία. Ναι, είναι συμβαστική τροπολογία, αλλά όχι με το oral amendment. Άρα λοιπόν, πρόεδρο, ποιο είναι υπέρ τη συμβαστική τροπολογία 36 χωρί το oral amendment, χωρί την ε, προφορητή τροποποίηση. Ναι, όταν μια πολιτική ομάδα είναι κατά του oral amendment, δεν περιλαμβάνεται στη συμβαστική τροπολογία του oral amendment. Άρα λοιπόν συμβαστική τροπολογία χωρί το oral amendment υπέρ. Κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Περνάμε στη 511, τροπολογία 511. Ψήφι υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία λοιπόν. Απορρίπτεται λοιπόν με 36 ψήφους κατά και 30 υπέρ. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 37 ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ε, ζητείται από τον πρόεδρο να ελέγξει, αλλά λέει ότι όχι ήταν σαφές το αποτέλεσμα. 528 λοιπόν τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Ψήφι υπέρ λοιπόν. 528. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 529 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 530 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. απορρίπτεται με 37 ψήφους κατά και 28 υπέρ. 531 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 532 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 533 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 534 ψήφι υπέρ, κατά εποχές ελέγχουμε 534 λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 35 ψήφους υπέρ και 30 κατά 535 ψήφοι υπέρ ψήφοι κατά αποχές ελέγχουμε αν και νομίζω ότι εγκρίνεται. Λήξη της ψηφοφορίας. 37 ψήφοι υπέρ, 29 κατά, εγκρίνεται. Εδώ έχουμε εκείνη η τροπολογία λοιπόν. Επόμενη ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν ενωθεί οι Έλληνες από όλες τις πολιτικές ομάδες. Έτσι έπρεπε να λέγεται αυτή η τροπολογία, λέει ο πρόεδρος. Άρα λοιπόν 38 ψήφοι υπέρ 29 κατά, άρα εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 3 και 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10, 11, 12. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε Λήξη της ψηφοφορίας. with the help of Mr. Karas. ψήφισε υπέρ τροπολογία. Κλείσαμε με αυτήν. Περνάμε στην 1622 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 νομίζω πως έχει καταπίψει. Οπότε 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές Ελέγχουμε. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 26 ψήφους υπέρ και 35 κατά. 25 τώρα υπέρ. Α, όχι. Συμβαστική τροπολογία 2 διορθώνει ο πρόεδρος. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 25 ψήφι ΠΕΡ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αλλά ας ελέγξουμε. Λήξη της υποφοριας 39 ψήφι υπέρ, 20 κατά. 37 ψήφι ΠΕΡ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 50. Α, όχι. Όχι, 36 διορθώνει ο πρόεδρος. Ψήφι υπέρ. Όχι τελικά. Τροπολογία, συγγνώμη, 36 υπέρ. Κύριε Πρέντα, νομίζω πως το διευκρινίσαμε αυτό στην αρχή της συνεδρίασής μας, ότι δηλαδή έχει αναλυφθεί από την άλλη πολιτική ομάδα αυτή η τροπολογία. Γι' αυτό και την ψηφίζουμε. 36 λοιπόν ψήφι Κατά. Θα ελέγξουμε. Die Ολοκληρώθηκε λοιπόν η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η τροπολογία με 36 ψήφου υπέρ και 29 κατά. 39 τώρα ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ελέγχουμε. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. 39 ψήφι υπέρ, 24 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 50 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 είναι η επόμενη που έχουμε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήταν σαφές αλλά μου ζητούν να ελέγξω. Λήξη της ψηφοφορίας. 30 ψήφοι υπέρ, 13 κατά, εγκρίνεται. 61 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ελέγχουμε. Πέραση της ψηφοφορίας. Οχτώ σαν δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Καλή σας μέρα. Ένα ξυπνήσω μερικούς. Ε, εντάξει, δεν περιμένω άλλο. Οι δύο τελευταίοι που απομένουν να ψηφίσουν Α συνεχίσουν να κοιμούνται. 31 λοιπόν, 31 ψήφοι υπέρ, 33 ψήφι κατά, άρα απορρίπτεται. 65 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 66 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 67 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ε, ψήφι υπέρ. Ελέγχουμε την 67 λέει ο πρόεδρος. Πέρας της ψηφοφορίας. 31 ψήφι υπέρ, 28 κατά εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 77. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. 42 ψήφι υπέρ, 24 κατά, εγκρίνεται. 74 ψήφι υπέρ, ε, συγγνώμη, 84 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 85 ψήφι κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 7 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 89 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 98 ψηφίπερ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε όμως. Λήξη της πληροφορίας. 53 ψηφίπερ 11 κατά οριακά εγκρίθηκε. Αστείευεται ο Πρόεδρος. Και περνάμε στην ψηφοφορία επί του συνόλου. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία επί του συνόλου της έκθεσης. Πλασκάρας on top, σε την ψήφο του συναδέλφου Κάρας. 42 ψήφια. Ε, ε, ε, υπέρ 11 κατά 11 εποχές θα θερμάμαστε συγχαρητήρια στην εισηγήτρια.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 bitte sich auf den Weg zu machen. Σας ε, παρακαλώ να αποχωρήσετε όσοι θέλετε να αποχωρήσετε. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 10 της ημέρα σας διαταξής μας. Σε συνεργασία λοιπόν με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Ρωσία, τον Σταλφοκάρας, Κάρας, έχουμε αυτό το σημείο εδώ προς και χαίρομαι που καλωσορίζουμε, καλωσορίζουμε τον, ε, ε, εδώ τον ε, Τόμας Μαϊχάρντινγκ που είναι ο Γενικός Διευθυντής για τα ζητήματα Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας και τον συγχαίρω βέβαια για την ανάληψη των καθηκόντων του και αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την συνεργασία μας τα επόμενα χρόνια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τη δυνατότητα που μου δίνετε για να μιλήσω σε σχέση με τη συνεργασία της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεργασία αυτή είναι πολύ σημαντική και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που θα μου δώσετε την ευκαιρία να απαντήσω και σε ό,τι ερωτήσεις έχετε για τις σχέσεις αυτές. Κύριε και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, μια από τις ιδιαιτερότητες είναι ότι έχω την ευκαιρία να σας ενημερώσω για τις συζητήσεις του Συμβουλίου και για τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε επί τη ευκαιρία του Συμβουλίου αυτού. Αρχίζω όμως λέγοντας ότι αυτή την εβδομάδα είναι δύο χρόνια από τότε που έγινε η παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας που όπως γνωρίζετε δεν αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα το αποσαφηνίζουμε κάθε φορά στις δηλώσεις μας βάσει της πολιτικής της μη αναγνώρισης. Και έχουμε και δήλωση για αυτή τη βδομάδα για την επέτειο ενός έτους στις 18 του μηνός. Οι προκλήσεις είναι πολλές και η κατάσταση είναι δύσκολη όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Ρωσία. Μια άλλη πρόκληση είναι και η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία με την αποσταθεροποίηση και εξαιτία της Ρωσίας. Ένα κεντρικό ζήτημα και μεγάλη ανησυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία βέβαια έχει να προχωρήσει σε μέτρα για να εφαρμόσει τη συμφωνία του Μίνσκ. Επιπλέον η Ρωσία παίζει ένα ρόλο κλειδί, μια που είναι συμπρόεδρος του ISG και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και πρέπει να παίξει επικοδομητικό ρόλο για να υπάρχει σταθερότητα. Η ανακοίνωση χτες της απόσυρσης του στρατού της Ρωσίας δήλωση που έκανε ο πρόεδρος Πούτιν ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της βίας στη Συρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί όλος ιδιαιτέρως για τον περιορισμό των ελεύθερων φωνών στην Ρωσία και όσον αφορά τον περιορισμό του κράτους δικαίου. Ας θυμηθούμε την Άντια Σαφτσένκο, μία περίπτωση που υπογραμμίζει ακριβώς αυτό το φαινόμενο. Η κατάσταση λοιπόν είναι πιο δύσκολη μετά, όπως είπα, την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας και εξαιτία των διεθνούς συγκυρίας οι σχέσεις μας με τη Ρωσία έχουν ιδιαίτερη σημασία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα ήταν κάτι που το βλέπαμε να έρχεται εδώ και καιρό. Υπάρχουν οι πτήσεις transit, τα θέματα τα φυτογενομικά και είναι πράγματα τα οποία έχει θέσει και η Αυστριακή Προεδρία. Μην ξεχνάμε και την πετρελαϊκή κρίση. Όλα αυτά τα πλαίσια λοιπόν οδήγησαν χτέ το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να συζητήσει για πρώτη φορά συνολικά τις σχέσεις με την Ρωσία μετά από την προηγούμενη φορά που ήταν ένα χρόνο πριν. Βέβαια, στόχος δεν ήταν η ανάπτυξη νέας πολιτικής απέναντι στη Ρωσία. Η προσέγγισή μας για τη Ρωσία παραμένει ίδια. Ότι θέλουμε ανοιχτό διάλογο στα πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Double Track. Αυτό δεν αφισβητήθηκε και αποσαφηνίστηκε. Το θέμα ήταν οι σχέσεις με την Ρωσία γενικά και όχι οι κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, κάτι το οποίο θα εξεταστεί αργότερα. Έτσι επιβεβαιώσαμε την ε, ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και ακριβώς η ενότητα είναι η δύναμή μας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πέντε αρχές θελήσαμε να παρουσιάσουμε στις χώρες μέλη που ορίζουν τη σημερινή μας πολιτική. Επαναλαμβάνω ότι δεν πρόκειται για την ανάπτυξη της πολιτικής μας απέναντι στη Ρωσία στο μέλλον, πρόκειται για το πλαίσιο μέσα στο οποίο σήμερα λειτουργούμε. Αυτές οι πέντε αρχές που δημοσιοποίησε μετά και εκπρόσωπος και που έγιναν απαιδεκτές από όλες τις χώρες ε, μέλη ομόφων είναι εξή. Πρώτον, πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ αποτελεί στοιχείο κλειδί για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στις σχέσεις μας. Δεύτερη αρχή, πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις με τους εταίρους μας ε, στα ανατολικά μας και με τους εταίρους μας στην Κεντρική Ασία και άλλους. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση για το πώς μπορεί να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η σχέση αυτή. Και θα συνεχίσουμε να συζητάμε για τις σχέσεις μας με τους εταίρους μας ανατολικά και στο επόμενο Συμβούλιο. Τρίτον, ενίσχυση της αντοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο για την ασφάλεια με τη στενή έννοια του όρου, μιλάμε και για θέματα όπως είναι ενεργειακή ασφάλεια, οι διάφορες απειλές στον κυβερνοχώρο, αλλά και άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και για την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση από πλευράς της Ρωσίας. Κάτι άλλο στο οποίο συμφώνησαν οι Υπουργοί είναι ότι ότι πρέπει να δούμε πώς εμπλέκεται η Ρωσία επιλεκτικά σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που είχαμε τον τελευταίο καιρό. Η Ιράν, η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, TPK, αντιτρομοκρατικές δράσεις, κλιματική αλλαγή, αλλά και άλλοι τομείς όπου σαφώς και υπάρχει εμπλεκόμενο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, πέμπτη αρχή. που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή σας, είναι η επιθυμία μας να στηρίξουμε περισσότερο την κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία και να επενδύσουμε σε επαφές με τον κόσμο και σε πολιτικές που έχουν να κάνουν με τον τομέα αυτό και διατήρηση βέβαια του διαλόγου με την επόμενη γενιά, με τους νέους της Ρωσίας, εκπαίδευση κλπ. Αυτές λοιπόν είναι οι πέντε αρχές γύρω από τις οποίες ε, συζήτησαν και αποφάσισαν ομόφωνα οι Υπουργοί χτες. Είναι ένα μήνυμα ενότητας που στέλνουμε δηλαδή και βάσει αυτών των αρχών θέλουμε και μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τη Ρωσία ακόμα και κάτω από αυτές τις δύσκολες ε, συνθήκες τις οποίες βρισκόμαστε σήμερα. Ευχαρίστω Πρόεδρε να επεκταθώ περισσότερο σε μία την άλλη από αυτές τις αρχές εφόσον το επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ο κύριος Κάρας έχει το λόγο τώρα. Κύριε Πρόεδρε και κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την ε, παρουσίαση. Γνωρίζετε ε, προφανώς ε, ότι εμείς χαιρετίζουμε την σαφήνεια αυτή τη έκθεση, αλλά α, μας δίνει και κάποιες ενδείξεις σε ό,τι αφορά δηλαδή την ανάγκη για την εντατικοποίηση του διαλόγου μας και σε σχέση με το πώς μπορούμε να οργανώσουμε αυτόν τον ε, διαλόγο. Ταυτόχρονα όμως θέτει ε, και το ζήτημα της μη ε, πλήρους των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη Συμφωνία του Μίντ και του τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο συνεργασίας με τα μέλη της Ντούμα και της Κάτω Βουλής της Ρωσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τίποτα καινούριο πάντως μετά την χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου. Αναφερθήκατε εσείς σε μία σειρά από πρωτοβουλίες. Η τέταρτη αποτελεί καινοτομία, η πέμπτη, τίποτα το καινούριο ουσιαστικά μας λέτε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τις διαπροσωπικές σχέσεις, ε, να έρθουμε σε επαφή με την ρωσική κοινωνία. Όσον αφορά την τέταρτη αρχή, αυτή είναι λίγο ασαφής για μένα. Κύριε Χάρτινγκ, θεωρώ ότι η Ρωσία ακολουθεί μια συγκεκριμένη στρατηγική, πολύ πιστά. Δυστυχώς όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απλώς κάποια συμφέροντα. Και πολλές φορές ενδιαφέροντα συμφέροντα θα έλεγα. που δεν προωθούνται πάντα επαρκώς ή πάρα πολύ προδήλως αν θέλετε, ιδίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Πάντως δεν βλέπω καμία στρατηγική τροποποίηση στη στάση της Ρωσίας. Υπάρχει κάτι τόσο το πολύπλοκο συμφωνία του Μίνσκ που δεν μπορεί να καταλάβει η ρωσική πλευρά. Τι ακριβώς πρέπει περαιτέρω να εξηγήσουμε στους Ρώσους προκειμένου να εφαρμόσουν αυτή τη συμφωνία. Και ξέρω ότι κάποιες αντιπροσωπείες βιάζουν να επισκεφθούν τη Μόσχα, αλλά από την άλλη οι Ρώσοι δεν αλλάζουν καθόλου τη στάση τους. Εξακολουθούν και έχουν τον μαύρο κατάλογο και όλες τις υπόλοιπες αρνητικές κυρώσεις κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς ποια αλλαγή πραγματικά βλέπετε αυτή τη στιγμή στη ρωσική στάση που θα μπορούσε όντως να μας οδηγήσει σε αυτό το οποίο είπατε, το selective engagement, το να καταφέρουμε να δεσπευτούμε επιλεκτικά σε κάποιους τομείς και να ενισχύσουμε το διάλογο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έγγραφα τα οποία έχουν εγκριθεί από κοινού, έχουν υπογραφεί, πρέπει πρώτα απ' όλα να εφαρμοστούν προκειμένου να διηγηθούμε στο μέλλον σε κάποιες αλλαγές. Αυτό αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Και εγώ δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σπουδαία νέα από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να μας ενημερώσετε δυνατόν για το τι εννοεί το Συμβούλιο όταν λέει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με την Κεντρική Ασία. Αν πραγματικά υπάρχει ένα περιθώριο για επιλεκτική δέσμευση και συνεργασία με τη Ρωσία, τότε μπορούμε να έχουμε selective engagement με περισσότερες περιοχές της Κεντρικής Ασίας. Βέβαια, υπάρχουν ορισμένες χώρες με τις οποίες δεν θα ήθελα να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με την μεταξύ αυτών των κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε απλώς να δεσμευθούμε με την περιοχή αυτή χωρίς να θέσουμε κάποιες προϋποθέσεις, χωρίς να τονίσουμε ότι υπάρχει επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε ποια διαδικασία προτίθεται να ακολουθήσει, να το Συμβούλιο προκειμένου να ενδυναμώσει τις σχέσεις του με την Κεντρική Ασία όπως λέει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε για την αρχή σε αυτή παρουσίαση όσον αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας και όσον αφορά τις πέντε αυτές βασικές αρχές στις οποίες αναφερθήκατε. Νομίζω ότι το πιο ουσιαστικό αυτή τη στιγμή είναι να εφαρμόζουμε αυτά για τα οποία δεσμευόμαστε. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνεπείς ως προς αυτό. Φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, διάφορα υπόγεια κινήματα, θα έλεγα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ουσιαστικά αποδυναμώνουν τη στάση την οποία θα έπρεπε να έχουμε απέναντι στη Ρωσία. Το να είμαστε σε επαφές με τους υπερμάχους της δημοκρατίας στη Ρωσία, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί όμως λένε ότι θα πρέπει οι κυρώσεις αυτές να στρέφονται κυρίως εναντίον των ατόμων εκείνων που βρίσκονται στον πιο στενό κύκλο του Βλαντιμίρ Πούτιν και να μην στρέφονται οι κυρώσεις αυτές εναντίον των περιοχών εκείνων στις οποίες υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι τελικά θα μπορούσαν να υποφέρουν εξαιτία των κυρώσεων αυτών. Βλέποντας συμπεράσματα του Συμβουλίου, βλέπω ότι παραμένουμε ενωμένοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση στη στάση μας. Ωστόσο το τίμημα της ε, ενιαίας αυτής στάσης είναι πάρα πολύ υψηλό. Και το λέω αυτό διότι επί του παρόντος προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική λύση η οποία ουσιαστικά παρουσιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα εξασθενημένη. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά κρίμα και λυπηρό να καταλήγουμε σε κάτι τέτοιο. Ιδίως αν δούμε το παρελθόν μας και το παρελθόν των σχέσεών μας με τη Ρωσία. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αντιμετωπίζουμε χώρες σαν τη Ρωσία με έναν τρόπο τόσο μη αποφασιστικό τελικά. Βλέπετε ότι η χώρα αυτή δεν ακολουθεί το κράτος του δικαίου και το έχει κάνει αυτό επανειλημμένος. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον τα όσα αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν στις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Πιστεύω πραγματικά, θέλω να ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία και ότι θα καταφέρουμε να παραμείνουμε ενωμένοι. Για Κονσάρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας δώσατε. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, αναλύοντας τη σημερινή κατάσταση της ε, Ρωσίας ως προς ε, την, οικονομική της δηλαδή κατάσταση, αν έχετε αναλογιστεί ποιες είναι τόσες αυτές για την Ευρώπη και για την Κεντρική Ασία. Ποια είναι δηλαδή τα συμπεράσματα που θα πρέπει να λύσουμε από την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία. Μήπως δηλαδή θα πρέπει να ασκήσουμε κριτική στον εαυτό μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα ε, μου θυμίζει λίγο μια προσέγγιση νηπιαγωγείου. Δηλαδή εμείς λέμε ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα αν δεν ε, τηρήσουν τα όσα έχουν ε, συμφωνηθεί στο πλήσιο της συμφωνίας του Μίτσικα. και από την άλλη πλευρά εκείνοι μας λένε ότι εμείς είμαστε μια χαρά, δεν πειράζει, επιβάλλεται μας κυρώσεις. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο δεν επιτυχάνουμε τίποτα σε βάθος χρόνου. Πώς λοιπόν, ρωτάω, μπορούμε να βρούμε ένα νέο τρόπο, μια νέα έναρξη εδώ, επανέναρξη του διαλόγου. Ich habe Fragen zu drei der... Ναι, θα ήθελα να θέσω ε, ερωτήματα σε σχέση με τρεις αρχές. Καταρχήν σε ό,τι αφορά την πρώτη αρχή. Ποια είναι η συζήτηση που λαμβάνει η χώρα στο επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών. Γιατί ο Υπουργό Εξωτερικών τη Γερμανία έχει την τάση να μιλάει για το Μίνσκ σαν να είναι και οι δύο πλευρές ε, εδώ της ε, σύραξη τη ε, της διένεξης που απορρίπτουν αυτήν την την, την, την επίλυση ε, του, του ζητήματος και αυτό γιατί για παράδειγμα με βάση τις εκθέσεις του ΩΣΑ βλέπουμε ότι ε, το LNR και άλλες ε, ομάδες είναι εκείνες που απορρίπτουν την όλη προσέγγιση άρα λοιπόν δεν βλέπουμε με αντικειμενικό τρόπο τη στάση της Ρωσίας οπότε θα ήθελα να ακούσω τι συζητάτε σε επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών και στο Συμβούλιο. Επίσης σε ό,τι αφορά τις υπηρετικές απειλές, τα hybrid threats θα ήθελα να ακούσω ποια είναι ε, στάση που υιοθετείται ε, για παράδειγμα και από την ε, Ηνωμένο Βασίλειο ή τις κάτω χώρες έναντι της Ρωσίας και θα ήθελα να ακούσω και τι σημαίνει αυτή η επιλεκτική εμπλοκή με τη Ρωσία, η επαφή με τη Ρωσία σε ό,τι αφορά ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι δηλαδή τα κράτη-μέλη εκείνα που θα ήθελαν να προωθήσουν τα συμφέροντά τους έναντι της Ρωσίας χωρίς να ε, τηρεί εκείνη τα όσα έχουν συμφωνηθεί στο Μίτσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Βάγκλε. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Έχουμε συναντηθεί στη Βιέννη αρκετέ φορές. Θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο ήταν σαφές στη συνάντηση ότι Διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν τη δικιά τους πορεία και τα δικά τους συμφέροντα όταν πρόκειται για τις σχέσεις με τη Ρωσία. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη στρατηγική όσον αφορά τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Δεύτερον, θέλω να γνωρίζω κατά πόσο κάποιος είπε πως το εμπάργκο ε, με τη Ρωσία ζημιώνει σημαντικά τα ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα στο σύνολό τους, αλλά και πιο συγκεκριμένα για διάφορες χώρες, η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή εξαιτίας αυτού του εμπάργου. Τέλος, αναφερόμαστε στη συμφωνία του Μίνσκ. Πολλοί σας ρώτησαν για αυτή τη συμφωνία και η ομάδα Μίνσκ που δημιουργήθηκε προκειμένου να λυθεί το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ και όπου εγκατέλειψε την έδρα της Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ της Γαλλίας, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος Στέτινα. Κύριε Χάρντινγκ, δύο ερωτήσεις έχω για σας. Πρώτον, το πρώτο που αναφέρατε κι εσείς, οι συμφωνίες δηλαδή του Μίνσκ, οι συμφωνίες αυτές δεν εφαρμόζονται, είτε πρόκειται για την κατάπαυση πυρός, είτε για άλλα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, τη Δευτέρα υπήρξε κανένα σημάδι για ένα σχέδιο Β, αντί για τις συμφωνίες Μίνσκ, αν δηλαδή έχουν οι συμφωνίες αυτές. Κάτι το οποίο είναι πιθανό να συμβεί. Και όταν μιλάω για σχέδιο Β, αναρωτιέμαι κατά πόσο σκεφτήκαμε να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αντιμετωπίσει κάποια επίθεση. Και επαναλαμβάνω κάτι που έχω πει ξανά και ξανά. Έχουμε σκεφτεί στρατιωτική τεχνολογία να την προσφέρουμε στην Ουκρανία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια ρωσική επίθεση. Υπάρχει λοιπόν εναλλακτικό σχέδιο αν δεν πετύχουν οι συμφωνίες του Μίνσκ. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερον, Γι' αυτά που είπατε για ευρυδικό πόλεμο και για παραπληροφόρηση από πλευρά της Ρωσίας. Θέλω να τονίσω εδώ ότι η άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ αδύναμη, υπερβολικά, θλιβερά αδύναμη. Η κυρία Μογκερίνη μετά από τις οδηγίες του Συμβουλίου έφτιαξε μια ομάδα για να αντιμετωπίσει τη ρωσική προπαγάνδα. Η ομάδα αυτή αποτελείται από 8 άτομα όλα και όλα. Και η κυρία Μογκερίνη δεν μπόρεσε να πετύχει ειδικά κονδύλια χρηματοδότηση. Αναγκάζεται να δουλέψει βάση του προπολογισμού που είχαμε έτσι καλλιώς μέχρι τώρα. Μα πώς θα αντιμετωπίσουμε έτσι τη ρωσική προπαγάνδα. Έχετε τίποτα συγκεκριμένες προτάσεις για να αντιμετωπιστεί αυτή η μαζική παραπληροφόρηση από πλευράς της Ρωσίας που κάνει τόσο μεγάλη ζημιά στις ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστώ. Επόμενος μιλητής. Δύο σχόλια ερωτήσεις έχω. Πρώτον, πολύ συχνά πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί με εκπλήσονται από αυτά που κάνει η Ρωσία το 2008 στην Γεωργία, στην Κρυμαία και την Ανατολική Ουκρανία στη συνέχεια και μετά πολλοί εξεπλάγησαν όταν η Ρωσία μπήκε στη Συρία. Χτες είχαμε τα νέα ότι αποσύρει τα στρατεύματά της η Ρωσία από τη Συρία. Οπότε ρωτάω πώς αναλύει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την κατάσταση και τι προβλέπει για το μέλλον, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα αν κάνει κάτι άλλο η Ρωσία, πρέπει να ξέρουμε πώς θα απαντήσουμε. Δεύτερον, όπως γνωρίζετε, υπάρχει η πρόταση πάνω από πέντε ευρωβουλευτών, αλλά και από εθνικά κοινοβούλια ευρωπαϊκών χωρών, για να αποφασίσουμε κυρώσεις κατά εκείνων που έχουν ευθύνες για την περίπτωση Σασένσκο. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Κομισιόν προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις σε συγκεκριμένα άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την κατάσταση και για τα ό,τι συνέβησαν με τη Σασένσκο. Κύριε Πρέσβη, ο κύριος Συμφωνώ με τις ερωτήσεις των προλαλισσάντων και θέλω να ξέρω κι εγώ τι συμπεράσματα βγάζουμε από άλλες παραβιάσεις της Ρωσίας. Διότι πρέπει να προλαμβάνουμε τα πράγματα και όχι να αντιδρούμε κατόπιν εορτής. Η δύναμη η ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από την ενότητά της. Οι αρχές που παραβιάζει η Ρωσία συνεπώς πρέπει να αναλυθούν. Ακριβώς αυτό που κάνει η Ρωσία είναι ότι παίζει με την ε, αναποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζει ότι θα βαρεθούμε, θα κουραστούμε και ότι θα αναγκαστούμε να κάνουμε συμβιβασμούς πάνω στις αρχές μας και τις αξίες μας. Αυτό είναι κάτι επικίνδυνο όμως όσον αφορά την μακρόπνοια στρατηγική μας. Ο δισταγμός δηλαδή η προσπάθεια επίτευξης συμβιβασμών είναι μια δυναμία από την πλευρά μας. Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή μας στο θέμα των στοχευμένων κυρώσεων απέναντι σε συγκεκριμένα άτομα. γίνεται με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε μέσω αυτών τη συμπεριφορά της Ρωσίας. Οι υπεύθυνοι για τη σύλληψη, την κράτηση της κυρίας Σατσένσκο νομίζω ότι πρέπει να τιμωρηθούν επίσης. Να τους επιβληθούν κυρώσεις δηλαδή. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής. Ο κύριος Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα συμπροσυπογράψω ε, και εγώ το ερώτημα που έθεσε ο συνάδελφος ό,τι αφορά το πώς μπορούμε να βρούμε έναν νέο τρόπο να αντιμετωπίσουμε, ε, να συνδιαλλαγούμε με τη Ρωσία. Ε, ο λόγος για τον οποίο για τον οποίο πήρα το λόγο είναι η χρήση ε, της λέξης νηπιαγωγείο από την πλευρά της Και αυτό γιατί. Η... Το να έχει κανείς να κάνει με το καθεστώς ε, του Πούντεν είναι καθόλου από το... το να έχει να κάνει κανείς ε, με ένα νηπιαγωγείο. Δηλαδή πρέπει να πω ότι ελπίζω ότι Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δεν ε, πρόκειται να αλλάξει τη στρατηγική που ακολουθεί τώρα, την ευρεία τη στρατηγική και την ανάλυση της, σκεπτόμενη ότι θα ήταν ε, καλό να προβούμε σε ένα διάλογο απλώς και μόνο για να υπάρξει ένας διάλογος με το καθεστώς της Μόσχας. Και θα ήθελα εδώ να ε, αναφερθώ και στα όσα είπε ο συνάδελφος ό,τι αφορά την έκπληξή μας με τα όσα έχουν συμβεί ξανά και ξανά σε σχέση με τη Ρωσία. Δεν θα πρέπει δηλαδή να είναι το σκεπτικό μας ότι μετά από την εγκληματική ε, προσχώρηση στη Ρωσία της ε, Κρυμαίας η Ρωσία βρίσκεται τώρα ε, ενώπιον ενός νέου κεφαλαίου που ανοίγει ε, σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές της σχέσεις. Δύο χρόνια λοιπόν μετά από την Κρυμαία ακούμε τώρα ειδήσει σε σχέση με την υποτιθέμενη απόσυρση ε, της Ρωσίας από τη Συρία. Δεν είναι δηλαδή, σύμπτωση αυτό ότι λίγες μέρες πριν από την δεύτερη επέτειο από την ε, Κρυμαία να ακούμε για αυτή την απόσυρση. Άρα λοιπόν εμείς που είμαστε και δεν θα πρέπει να είμαστε αφελείς και σίγουρα δεν θα κερδίσουμε τίποτα από έναν διάλογο με τη Ρωσία ο οποίος απλά διεξάγεται για χάρη του διαλόγου και δεν έχει καμία σκοπιμότητα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ακούστηκαν πάρα πολλά ερωτήματα, οπότε θα προσπαθήσω να απαντήσω στα περισσότερα από αυτά και στα σχόλια που έγιναν. Καταρχής καταρχήν να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Κάποια μέλη αυτής της ε, Επιτροπής ανέφεραν ότι εξεπλάγησαν από το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ε, κάποιες ιδέες ε, σχετική εκδήλωση. Αλλά όπως σας είπα ο στόχος της, ε, ε, της χθεσινής ε, συνάντησης δεν ήταν να υπάρξει μια νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Ρωσίας, αλλά ήταν αντιθέτως να υπάρξει μια ενότητα σε ό,τι αφορά δηλαδή την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με κάποιες βασικές αρχές και οι οποίες αρχές θα αποτελέσουν το βασικό άξονα για την περαιτέρω δράση μας. Οπότε με βάση και τα σχόλια που άκουσα σήμερα εδώ ε, καταδεικνύεται ότι ακριβώς είναι δύσκολο να βρούμε ενότητα, ένα κοινό μέτωπο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Ρωσίας και νομίζω πως αυτό που πετύχαμε χθες ήταν ακριβώς αυτό και είναι σημαντικό ότι δηλαδή μπορούσαμε να, μπορέσαμε να βρούμε μια ενότητα και να ε, ε, τονίσουμε την ενότητα μεταξύ μας έναντι της Ρουσίας και νομίζω πως καμία, ε, κανένας από τους συμμετέχοντες δεν εξέφρασε την αντίρρησή του απέναντι σε αυτές τις γενικές αρχές που καθορίσαμε χθε. Επίσης, εγώ δεν είμαι κάποιος ο οποίος υποτιμά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τη σήμερα ημέρα σε σχέση με το ζήτημα της Ρωσίας. Ως ε, νεαρός ε, σχετικά αυστριακός διπλωμάτης είχα υπηρετήσει στην ονομαζόμενη τότε Εσουσουδού στα τέλη της δεκαετίας του 90, δηλαδή υπήρξε τότε μια μεγάλη ελπίδα για αυτή τη χώρα σε σχέση με τα όσα βιώνουμε σήμερα και νομίζω πως είχα, ε, θυμάμαι πως είχα συναντηθεί τότε ε, με τον κύριο Φανάσεφ ο οποίος ήταν δηλαδή ο τριτή του κινήματος Memorial και ο οποίος ήταν διατεθειμένος ε, να συζητήσει για πρώτη φορά δημοσίως τα εγκλήματα της ελληνικής περίοδου και όλα αυτά μας εκπλήσουν δηλαδή σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν σήμερα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει σήμερα τι σήμαινε ε, τότε στην περίοδο του Στάλιν ε, το να είναι κανείς ξένος πράκτορας και αποτελεί πραγματικά έκπληξη το γεγονό ότι αυτή, αυτό το κίνημα με Memorial αποκαλείται σήμερα από το Moodle ως ε, ελεγχόμενο από τους ξένους όργανο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και στο πλαίσιο της πρόθεσης της κοινωνίας των πολιτών και νομίζω πως και το Συμβούλιο γνωρίζει καλά το τι συμβαίνει σε αυτό το επίπεδο στη Ρωσία. Ένα ακόμα σχόλιο που θα ήθελα να κάνω γιατί τέθηκαν και ερωτήματα ε, σε ό,τι αφορά το ρόλο του σχετικού φορέα. Ε, δεν ε, αναφέρθηκε το ζήτημα των, της δόμησης, αν θέλετε, της διάθρωσης των σχέσεων μας με τη Ρωσία, γιατί κάθε φορά που έχουμε συναντήσεις με τη Ρωσία, ε, τίθεται ε, ξανά και ξανά το ερώτημα ότι έχουμε αυτέ τι δύο συνόδου κορυφή. Δεν θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε αυτέ τι συνόδου ε, και να τι χρησιμοποιήσουμε για αυτό το λόγο. Θα πρέπει να πούμε ότι, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το μόνιμο Συμβούλιο Εταιρικέ Σχέσει, να πούμε ότι έχει ήδη διαλυθεί γιατί θεωρήθηκε ότι αυτό το συγκεκριμένο όργανο δεν ήταν κατάλληλο για τι σχετικέ επαφέ με τη Ρωσία. Σε ό,τι αφορά τι τις επιλεκτικές σχέσεις, το selective engagement όπως αναφέρεται σε σχέση με τη Ρωσία, θα πρέπει να πω ότι δεν είναι κάτι το καινούριο. Δηλαδή, οι γενικά οι σχέσεις στη διεθνή σκηνή με τη Ρωσία είναι κάτι το δύσκολο για μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν Νομίζω πως ε, χρειάζεται κάποιος να είναι προφήτης για να προβλέψει ότι και, μέσα στο, και στο μέλλον θα συνεχίσουν να είναι αυτές δύσκολες οι επαφές με τη Ρωσία. Ωστόσο, για ζητήματα όπου έχουμε ένα συμφέρον να έρθουμε σε επαφή με τη Ρωσία, είναι σημαντικό και νομίζω πως το Ιράν αποτέλεσε ένα σαφές ε, παράδειγμα ότι είχαμε ακριβώς αυτή την επιλεκτική επαφή και τον επιλεκτικό διάλογο με το Ιράν. Ε, και νομίζω πως και σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας στη Συρία είναι σημαντικό να ξεκινήσει ένα διάλογο σε ό,τι αφορά το ρόλο τη Ρωσία στη Συρία. Και νομίζω πω ε, αυτό ο διάλογο θα ήταν προ όφελο, προ το συμφέρον ε, ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα δε για τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία είναι τα πλέον εκτεθειμένα στην εξωτερική πολιτική τη ε, Ρωσίας για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τους φυτιογενομικούς ελέγχους. Ε, να πούμε ότι η Ρωσία, παρότι ακούγεται πολύ τεχνικό αυτό το μέτρο, ε, η Ρωσία χρησιμοποιεί λοιπόν αυτούς τους φυτιογενομικούς ελέγχους για να διαχωρίζει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή εφαρμόζει με διαφορετικό τρόπο αυτούς τους κανόνες σε κάποια κράτη-μέλη και με διαφορετικό τρόπο σε άλλα. Άρα λοιπόν έχει νόημα το να προβαίνουμε σε αυτό το selective engagement, σε αυτή την επιλεκτική επαφή με τη Ρωσία, γιατί μόνο ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακριβώς μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, θεσμικών της εκπροσώπων μπορεί πράγματι να επιδείξει ένα κοινό μέτωπο εναντί της Ρωσίας, να μιλήσει δηλαδή με μια ε, φωνή. Άρα λοιπόν δεν αποτελεί κάτι το καινούριο αυτή η επιλεκτική προσέγγιση της Ρωσίας. Το κάνουμε ήδη, το πράττουμε ε, σε σχέση με κάποια ζητήματα σε σχέση με τη Ρωσία. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία του Μίνσκ, ήταν σαφές χθε και συζητήθηκε από του υπουργού ότι η για να υπάρξει κάποια οποιαδήποτε βασική αλλαγή σε σχέση μας με τη Ρωσία θα πρέπει ε, να ε, ισχύσει η προϋπόθεση της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας των ε, όσων προβλέπει η συμφωνία του Μάσκ. Προφανώ ε, και οι δύο πλευρές δεσμεύονται από αυτή τη συμφωνία, δηλαδή και η Ρωσία και η Ουκρανία και εμείς επιμένουμε απέναντι στην Ουκρανία ότι θα πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από τη δική τη πλευρά. Ωστόσο γνωρίζουμε ταυτόχρονα και ποιε είναι οι δυσκολίε στα ανατολικά αυτή τη Δηλαδή η παρουσία του ΩΣΑ σε, σε όλες αυτές τις περιοχές είναι πολύ δύσκολο να ε, ε καταλήξουν τελικά οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία για τα εν λόγω ζητήματα. Άρα λοιπόν και εδώ η εικόνα ε, διαμορφώνεται και σε μεγάλο βαθμό και διέπεται σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση της ε, ασφάλειας, της υποχρεώσει ασφάλεια στα ανατολικά τη χώρα. και εδώ βέβαια ε, έχει μεγάλη ευθύνη γι' αυτό η Ρωσία ακριβώς επειδή δεν ε, πληρεί τι ειδικέ τη υποχρεώσει που πηγάζουν από τη Συμφωνία του Μίνσκ. Και προφανώς η ε, φωνή της Γερμανίας και της ε, Γαλλίας ε, έχουν πολύ ιδιαίτερο ειδικό βάρος στο πλαίσιο για τις διαδικασίες της Νορμανδίας. Επίσης μου τέθηκε μια ερώτηση ό,τι αφορά την ομάδα του Μίνσκ. Όπως γνωρίζετε η μετεκπρόσωπος επισκέφθηκε πρόσφατα το Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία και κατέστησε πολύ σαφές στο πλαίσιο αυτών των επισκέψεών της ότι υποστηρίζουμε πλήρως από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προτάσεις των συμπροέδρων της Επιτροπής του Μίνσκ, όπως δηλαδή αυτές ε, αποκρισταλώνονται και στις ε, ε, σχετικές αρχές. Και θεωρώ πως σε ό,τι αφορά τη δική μα στάση απέναντι στη συμφωνία του Μίνσκ, θεωρούμε πω θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρω και σε σχέση με αυτό υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών και των Υπουργών, ότι δηλαδή μόνο πολιτικής φύσης μπορεί να είναι η λύση που θα δοθεί σε αυτήν την, ε, στην επίλυση της πολύ δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζει η Ουκρανία τη σήμερα ημέρα στα ανατολικά της χώρας αυτής. Τώρα, κάποια, κράτη, ε, ε, κάποια μέλη εδώ της Επιτροπής ε, με ρώτησαν σε σχέση με τις ειδικές πληροφορίες που έρχονται από τη Ρωσία και το, το, Stratcom και το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Θεωρώ ναι πως θα πρέπει να ισχυθεί ε, περαιτέρω, αλλά από την άλλη πλευρά να πω ότι και οι Υπουργοί ήταν ε, πολύ θετικά διακείμενοι απέναντι δηλαδή στην περαιτέρω εξέλιξη αυτή του ρόλου της Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής δράση. Για πρώτη φορά υπάρχει μια τέτοια ε, δομή και νομίζω πως έχουμε προχωρήσει αρκετά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημα που μας τέθηκε, σε ό,τι αφορά δηλαδή το πώς ερμηνεύουμε εμείς την πλέον πρόσφατη απόφαση της Ρωσίας σε ό,τι αφορά την απόσυρση από τη Συρία, νομίζω πως είναι πολύ νωρίς για να δώσουμε εδώ μία οριστική απάντηση ως προς τι ακριβώς σημαίνει δηλαδή αυτή η κίνηση της ε, Ρωσίας στο γενικότερο ε, γεωπολιτικό πλαίσιο. Δηλαδή θα πρέπει να την αξιολογήσουμε αυτή την ε, κίνηση προσεκτικά και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά οποιοδήποτε βήμα γίνεται για την αποκλιμάκωση της βίας εντός της Συρίας και συμβάλλει στην πάυση των εχθροπραξιών αποτελεί σημαντική σημαντικό, σημαντικό βήμα για την ε, ειρηνευτική διαδικασία και ε, συμβάλλει ακριβώς στη διαδικασία εξέβρεσης ε, πολιτικής λύσης στον πόλεμο στη Συρία. Νομίζω πως είναι λίγο πρόωρο να πούμε ότι πράγματι γίνεται ένα τέτοιο βήμα και επιτυχάνουμε κάτι τέτοιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το, το ζήτημα των συμπληρωματικών listing, σε ό,τι αφορά την την ε, ιδιαίτερα δύσκολη ε, κατάσταση στην οποία αντιμετωπίζει η Νέντε Σαφτσέγκο, να πω ότι όποιο περαιτέρω ε, listing ε, γίνει θα πρέπει προφανώς να συμφωνηθεί στο επίπεδο του Συμβουλίου και το Συμβούλιο θα πρέπει να εξετάσει οποιαδήποτε τέτοια πρόταση με βάση τα νομικά ε, κριτήρια τα οποία έχει προβλέψει η σχετική νομική πράξη. Αυτά λοιπόν θα αποτελέσουν το κριτήριο για οποιοδήποτε listing αλλά σε ό,τι αφορά ειδικότερα την περίπτωση της Νάτια Σαφτσέγκο νομίζω πως θα είδατε την πολύ εμφατική δήλωση της εκπροσώπου για αυτό το ζήτημα και ασχολείται με αυτό προσωπικά και έχει καταστήσει σαφέστατο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεωρεί πως η απαγωγή της Νάντια από την Ουκρανία και η κράτησή της αποτελεί ε, παραβίαση των υποχρεώσεων σε επίπεδο του διεθνούς δικαίου της Ρωσίας σε ό,τι αφορά δηλαδή και το δικαίωμα για δίκαια ε, δίκη και θεωρεί πως οι τελευταίες, τα τελευταίες ειδήσει σε ό,τι αφορά την κατάσταση υγείας της κ. Σαφτσέγκο είναι πολύ κακές οπότε καλεί τη Ρωσία να απελευθερώσει για ανθρωπιστικού λόγου και χωρί προποθέσει την Αντία και εμεί ε, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε ε, πολύ προσεκτικά οποιαδήποτε συνέχεια δοθεί σε αυτήν την ε, δήλωση. Και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά το διάβημα αυτό με βάση δηλαδή και τη στάση που έχει οθετήσει η Ρωσία κατά τα τελευταία χρόνια, αλλά εμεί θα συνεχίσουμε να επιμένουμε σε αυτό το ζήτημα και επί του οποίου έχουμε ήδη εκφραστεί ε, με ενωμένο μέτωπο και με πολύ σαφή και κατηγορηματικό τρόπο. Ελέγχω, Πρόεδρε, αν εδώ στη λίστα μου αν έχω απαντήσει σε όλα τα σχόλια που μου απευθύνθηκαν. Ένα ζήτημα από το οποίο θα έπρεπε να είχα θέσει ευθύ εξ αρχή είναι ότι αυτές οι πέντε κατευθυντήρες, αν θέλετε, αρχές, οι βασικές αρχές, πάντοτε ισχύουν ε, υπό την επιφύλαξη και σεβόμενη την ε, ε, ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλεια και άμυνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό τονίστε και από την εκπρόσωπη και από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή αυτή η προσάρτηση της Κρυμαίας προφανώς αποτελεί παραβίαση της τάξης ασφαλείας στην Ευρώπη και θα συνεχίσουμε να το τονίζουμε αυτό και να το καθιστούμε σαφές στη ρωσική πλευρά και θα αποτελέσει τμήμα των, της ε, δραστηριοποίησή μας σε σχέση ε, με τη Ρωσία και νομίζω πως ε, θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα και εν του γενικότερου πλαισίου των οικονομικών κυρώσεων. Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία θίγονται περισσότερο από άλλα από αυτές τις οικονομικές κυρώσεις, αλλά πρόκειται για αποφάσεις επί της αρχής οι οποίες ελήφθησαν εν ώψη μιας κατάστασης η οποία δεν έχει βελτιωθεί μέχρι στιγμής. Και αυτό λοιπόν αναφέρθηκε για μία ακόμα φορά ε, από τους υπουργού ε, χθες ε, στο Συμβούλιο ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ προκειμένου για να υπάρξει μια αλλαγή της στάσης μας και βέβαια τον Ιούνιο θα υπάρξει και πάλι μια αναθεώρηση αυτή των κυρώσεων. Αυτά πρόεδρε θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες, για αυτήν την πολύ καλή συζήτηση που είχαμε. Προσβλέπουμε σε μια πολύ καλή συνεργασία εκ νέου στο μέλλον και σε ευχόμαστε καλή επιστροφή. Καλό ταξίδι. Äh, Τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξή μας είναι η εστίσταση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά την ε, σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο αγαπητός Άντρε Κόβατσεφ είναι ο εισηγητής μας για αυτή τη σύσταση. Όμως ε, πέρσι υπήρξε μια έκθεση πρωτοβουλίας για αυτό το ζήτημα, οπότε φέτος επιστρέφουμε και πάλι αν θέλετε ε, στην συνήθι μας πρακτική αν θέλετε, δηλαδή έχουμε σύσταση πλέον από την πλευρά του Κοινοβουλίου και πάλι έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, οι τροπολογίε θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι πότε, μέχρι Our proposal is that we have amendment time until Η Γραμματεία με ενημερώνει ότι η προθεσμία κατά την κατάσταση των τροπολογιών είναι 21η Μαρτίου, 12 ώρα. Ούτω ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε από εκεί και μετά. Αλλά κάποιος είδαμε εδώ, ήθελε αρχικά να προτείνει την 17η Μαρτίου. Γραμματεία είναι σύνδεση που προτείνει τέτοιου είδους προθεσμίες. Ότι δηλαδή επειδή όσοι καταθέτουν ε, τροπολογίες είναι πολύ απασχολημένοι, αν έχουν χρόνο για να εξετάσουν το email τους. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για όλες αυτές τις πληροφορίες που δώσατε. Στις δύο προηγούμενες νομοθετικές θητείες του Κοινοβουλίου ήταν ο κύριος Λάμστροφ, ο μόνιμος εισηγητής μας, το 2008 και το 2014 και κατάφερε να καταρτήσει 7 εκθέσεις όσον αφορά την σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Κάλυψε την περίοδο εκείνη κατά την οποία ήταν εισηγητής. Στην υφιστάμενη νομοθετική θητεία δεν είχαμε σύσταση για το 2014 και το 2015. Είχαμε κάποιες πιο γενικές εκθέσεις όσον αφορά την Ηνωμένα Έθνη. Ένας ακόμας λόγος για τον οποίο το Προεδρείο αποφάσισε να ξεκινήσει εκ νέου με την κατάρτιση συστάσεων είναι το ότι θέλουμε να αναζωογοποιήσουμε την ομάδα εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΗΕ καθότι αυξάνονται όλο και περισσότερο οι που έχουμε ω Κοινοβούλιο από αυτή την ομάδα εργασία. Κανονικά κάθε χρόνο, το Μάιο ή τον Ιούνιο, εγκρίνουμε κάποιες συστάσεις για την σύνοδο που λαμβάνει η χώρα το Σεπτέμβριο. Επομένως, θα πρέπει στην Ολομέλεια του Μαΐου να εγκριθούν οι συστάσεις αυτές και αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να ψηφίσουμε εδώ στην ΑΦΕ τον Απρίλιο. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, καταφέραμε με τη Γραμματεία να εξασφαλίσουμε μια παράταση της προθεσμίας κατάθεσης τροπολιών 21 Μαρτίου 12 το μεσημέρι. Σας ζητώ λοιπόν ή δυνατόν οι τροπολογίες σας να είναι γραμμένες στα αγγλικά, καθότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας μέχρι την ψηφοφορία που θα διεξαχθεί όπως σας είπα τον Απρίλιο. Έχετε στους φακέλους σας επίσης το σχέδιο εκθεσής μου το οποίο αναφέρεται σε οκτώ σημαντικούς τομείς, ειρήνη και ασφάλεια, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μη διάδοση και αφοπλισμός, μετανάστευση, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου, ανάπτυξη, κλιματική αλλαγή, Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταρρύθμιση του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, προβλέπονται και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν και αναφέρομαι βέβαια στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να δώσουμε και συνέχεια στην προηγούμενη έκθεση του κύριου Τέρου Ένινγκ καλύτερη ευθυγράμμιση επίσης της αντιμετώπισης των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες να μπορούν και αυτοί να καλυφθούν στην ανθρωπιστική δράση των Ηνωμένων Εθνών και επίσης να συμπεριλάβουμε επίσης και τις συστάσεις του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου του 2016 όσον αφορά την Μέση Ανατολή. Και να αναφερθούμε επίσης και στις ε, ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που γίνονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία. Προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές και με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων προκειμένου να καταλήξουμε σε μία ενιαία βάση συστάσεων και προσβλέπω στην περαιτέρω συμβολή που θα έχουν αυτοί οι σκιώδεις εισηγητές στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου συστάσεων. Κύριε Πρόεδρε που αποσιάζετε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω <laughs> τον λόγο στον αγαπητό συνάδελφο κύριο Παντσέρη, ο οποίος είναι σκιώδης εισηγητής για τους σοσιαλιστές μας. σε ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Παντσέρη. Δεν είμαι σκιώδης εισηγητής, αντικαθιστώ μάλλον τον σκιώδη εισηγητή, Σωράια Πόστο, ο οποίος ε, βρίσκεται στην Γενέβη για μια αποστολή του Κοινοβουλίου εκεί. Ο κύριος Πόστ λοιπόν θέλει να συγχαρεί τον ε, εισηγητή για αυτό το σχέδιο έκθεσης και προσβλέπει και αυτό σε μια περαιτέρω συνεργασία για την έκθεση αυτή, τονίζει ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάει με μια κοινή και νέα φωνή στα Ενωμένα Έθνη και να καταλήγει σε κοινό μέτωπο και κοινέ τοποθετήσει όσον αφορά τα ζητήματα με τα οποία ασχολούνται τα Ενωμένα Έθνη. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί μα βοηθά να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο σεβασμό του στα πλαίσια τη εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τροπολογίες που θα κατατεθούν από εμά θα έχουν να κάνουν με κάποια συγκεκριμένα κεφάλαια και με τους τίτλους των κεφαλαίων. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να βασιστούμε στους τρεις πυλώνες των εθνών, ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα, ασφάλεια και ανάπτυξη. Επομένως, θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο την ε, υιοθέτηση του ψηφίσματος 1325 και 2142 όσον αφορά την ειρήνη, την ασφάλεια και το ρόλο των γυναικών. Πρέπει επίσης να προωθήσουμε περισσότερο τα ψηφίσματα των ΗΕ... Εθνών για τους ανθρώπους που ανήκουν στην κοινότητα ΛΟΑΔΜΑ να προωθήσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να προσθέσουμε μια κάποια μνήμα όσον αφορά τους οργανισμούς εκείνους που εργάζονται για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να αναφερθούμε επίσης στην επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος, τη διένεξη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Φαντάζομαι όμως ότι θα προβλέψετε τον απαραίτητο χρόνο μαζί με τους κοιόδης συγητές, κύριε συγητά, προκειμένου να συμπεριλάβετε όλα αυτά τα επιπλέον σημεία στην έκθεσή σας. Uh, like to congratulate... Πρόεδρε, Ευχαριστώ. Συγχαίρω και εγώ τον εισηγητή, τον κύριο Κόβατσικ, για τις προσπάθειες του προκειμένου να ετοιμάσει αυτή την ισορροπημένη έκθεση. Πράγματι είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να τονίσει τις προτεραιότητές της εν ώψη της 71ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν πολλά παγκόσμια ζητήματα και οι συστάσεις μας θα ήταν μια ευκαιρία να δείξουμε στον κόσμο ολόκληρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μιλήσει με μία φωνή. Ως και εισηγητής από την ομάδα των φιλελευθέρων, θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πετύχει στις συστάσεις να συμπεριλαμβάνει και κάποιες σημαντικές προτάσεις υπέρ των αξιών μας. Να υπογραμμίζει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κλιματική αλλαγή, την ανάπτυξη και την πρόθεση του κράτους δικαίου. Αλλά θα ήθελα συγχρόνως να επιστήσω την προσοχή σας στο εξή. Προκειμένου να καταλήξουμε στον καλύτερο υποψήφιο για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα και τη δυνατότητα που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Στις συστάσεις λοιπόν θα ήθελα να συμπεριλάβουμε ότι θέλουμε μεταρρυθμίσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Αθηνών προκειμένου να καταπρίζει αυτό τη, καλύτερα την παγκόσμια πραγματικότητα και να μπορέσει καλύτερα να αντιμετωπίσει τις σημερινές και τις μελλοντικέ προκλήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ μιλάω εκ μέρου τη συναδέλφου τη κυρία Λόχμπιλερ, που θέλει να συγχαρεί και εκείνη τον εισηγητή για το εξαίρετο έργο του. Ω ομάδα, πολύ χαιρόμαστε που ακούμε την αναζωγόνηση του ΟΙΕ. Συμφωνούμε απόλυτα, ευχόμαστε κάθε επιτυχία και καλή δύναμη. Τρία σημεία θέλω να αναφέρω. Το πρώτο, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, έχει να κάνει με τη φετινή χρονιά όπου θα εκλεγεί ο νέος Γενικός Γραμματέας και ελπίζουμε να υπάρξουν και μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την εκλογή αυτή. Να προταθεί για παράδειγμα και μια γυναίκα υποψήφια έτσι για αλλαγή. Δεύτερον, στενομένα έθνη τη Γενική Συνέλευση μια νέα ομάδα εργασίας για τον αφοπλισμό δημιουργήθηκε. Ζητάμε λοιπόν από τις χώρες μέλη να στηρίξουν τις δραστηριότητε αυτές της νέας ομάδας εργασίας. Τέλος, έχουμε απογοητευτεί που οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν συνεισφέρει πιο συγκεκριμένα στις ειρηνευτικές αποστολές στο ΙΕ του 2015 με δυνάμεις. Είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ. ο κύριος Κόβατσεφ για να απαντήσει στα σχόλια για τις συστάσεις. Να πούμε κάτι ε, για υποψήφιους ε, στη θέση του Γενικού Γραμματέα, γυναίκες, τι λέτε. Ευχαριστώ. Κυρίως για το θέμα αυτό του φίλου, την ισορροπία δηλαδή μεταξύ των δύο φίλων, που, τώρα που έχουμε την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Είναι ένα σημαντικό κριτήριο η ισορροπία αυτή. Ευχαριστώ τους σκιώδεις εισηγητές για τα σχόλιά τους. Έτσι καλλιώς θα ξαναβρεθούμε και θα συζητήσουμε τροπολογίες. Σίγουρα επί τη ευκαιρία αυτή θα καταλήξουμε σε ένα καλό συμβιβασμό για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με μία φωνή πράγματι και να συστήσουμε στο Συμβούλιο να ακολουθήσει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμφωνώ για την ε, υψηλή αξία, για τις ειρηνευτικές δυνάμεις, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, κλιματική αλλαγή. Και όλα αυτά θα τα δεχτώ στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ.